Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση για να μην καθυστερήσουμε. Φτάνουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας της Επίτροπης από την ε, Κεντρική Υπηρεσία στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της. Έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Κάρελ Πρίνγκστεν, μέλος, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου από το 2006 και που είναι από το μήνα Απρίλιο ε, στο τρίτο σώμα. Ο κύριος Πρίνγκστεν υπήρξε ευρωβουλευτής και πολλές φορές υπουργό ε, στην βελγική κυβέρνηση. Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά κύριε Πρίνγκστεν και εξ ονόματος της Επιτροπής μας εφόσον την περασμένη εβδομάδα ακολουθώντας την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ενέκρινε την, τον διορισμό σας στο ελεγκτικό συνέδριο στο πνεύμα των αγαστής συνεργασίας με το ελεγκτικό συνέδριο, ο κύριος Πίνξτεν δέχτηκε την πρόσκλησή μας για να λάβει μέρος στην συζήτηση της έκθεσης 1 του 2011 του ελεγκτικού συνεδρίου για την αποκέντρωση της διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας τη Επιτροπής από την έδρα της στις αντιπροσωπείες. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε προς όφελος της Επιτροπής Ανάπτυξης που είναι η υπεύθυνη Επιτροπή για την έκθεση πρωτοβουλία Πρωτοβουλίας. Ο εισηγητός μας είναι ο κύριος Μαυρονικόλας. Σας προτείνω λοιπόν να κάνουμε σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σας προτείνω να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μαυρονικόλα και μετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πίγκστεν. Ο κύριος Μαυρονικόλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φίλιπ Κάσμαρεκ για την πρωτοβουλία του να συντάξει μια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από την έδρα της στις επιφορτισμένες αντιπροσωπείες της στην παράδοση βοηθείας. Στη συνέχεια θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Καρλ Πίξτεν, μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός για την προώθηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι προτεραιότητες της Ένωσης θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στα πλαίσια μιας ενισχυμένης ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλώντας για αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από την έδρα της στις επιφορτισμένες αντιπροσωπείες της, πρέπει να αναφέρω ότι η συναρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και Επιτροπής αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι στα θέματα προγραμματισμού αναπτυξιακής βοήθειας, ειδικά μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, κατά την οποία αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γι' αυτό άλλωστε πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των δύο προκειμένου να ισορροπήσει το σύστημα συναρμοδιότητας σε αναπτυξιακές δράσεις και να καταστεί πιο αποτελεσματικό. Επίσης, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία σε κατατόπους αντιπροσωπείες έχει συμβάλει στην βελτίωση ταχύτητας των δράσεων, στην ποιότητα της βοήθειας και στην πιο αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό έρχεται και το ζήτημα της κατανομής των ανθρωπίνων πόρων στις αντιπροσωπείες, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να τονιστεί στο σχέδιο έκθεσης. Συγκεκριμένα, το εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με την εξωτερική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί, αλλά να είναι και μόνιμο, ώστε να διατηρείται θεσμική μνήμη και μία συνέχεια στην ίδια την υπηρεσία. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε σχέση με την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης τεχνικών και οικονομικών ελέγχων και αξιολογήσεων στις αντιπροσωπείες. Όχι τόσο για το θέμα της διαχείρισης, αλλά περισσότερο για το θέμα της επίτευξης των στόχων. Είναι απαραίτητο για τις αντιπροσωπείες να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για την ολοκλήρωση του έργου τους με αποτελεσματικό τρόπο. Στο σημείο αυτό θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει ένα ανεπίσημο έγγραφο από αρκετά τα οποία ζητούν να έχουν μεγαλύτερο λόγο και ανάμειξη στον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Ράσης λόγω του ότι συμβάλλουν κατά το 1 τρίτο του προσωπικού της υπηρεσίας με εθνικούς διπλωμάτες. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πιστεύει πως οποιασδήποτε αλλαγές απαιτούνται στον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρέπει να γίνουν με πολλή προσοχή. Δεν θα θέλαμε να εθνικοποιηθεί η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προγραμματισμός των χρηματοδοτικών μέσων που αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ίσως να πρέπει να επανα... επανεξεταστεί. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης, ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο της γνωμοδότησης και να το εμπλουτίσουμε με περισσότερα στοιχεία όπου θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Επειδή στη σύνταξη της γνωμοδότησης υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του κειμένου, περισσότερα στοιχεία ίσως προσθεθούν μετά την κατάθεση τροπολογιών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως επίσης και τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη τους βοήθεια. Thank you. Merci. Je vais donner la... Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πίξτεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως υπενθυμίσατε και εσείς, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι όμως η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και σας την ίδια ως πρόεδρο, αλλά και τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την πρόσκλησή σας. Όπως δίχως όλο γνωρίζετε, το ελεγκτικό συνέδριο έρχεται συχνά εδώ και είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας αλλά και για σας να υπάρχει αυτή η επαφή, να ερχόμαστε δηλαδή στις ειδικέ επιτροπές. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σχετικά με το έγγραφο, της διαχείριση εξωτερικής ε, βοήθειας και την αποκέντρωση της βοήθειας αυτής. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή σας. Φυσικά και διάβασα το έγγραφο το οποίο εκείνο ετοίμασε και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το κείμενό του. Πραγματικά αντιλαμβάνεται την ε, ουσία και περιλαμβάνεται η ουσία ε, του ζητήματος το έγγραφο αυτό του εισηγητή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω μερικά λόγια για να πλαισιώσω λιγάκι το θέμα αυτό. Και μετά θα έρθω στον έλεγχο και τα ευρήματα του ελέγχου. Και θα τελειώσω με μερικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά λοιπόν αυτή τη διαδικασία αποκέντρωση, ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2004. Χρειάστηκαν δηλαδή δύο με τρία χρόνια προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή. Όπως δίχως άλλο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε ελέγχους. Το 2005 αλλά τα αποτελέσματα, τα ευρήματα είναι γενικά θετικά. Το 2005 βέβαια ήμασταν μόλις αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας, οπότε ήταν κάπως νωρίς να αξιολογήσουμε πραγματικά τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό και το 2009 στο σώμα αριθμός 3, ονομάζουμε, πριν ονομαζόταν Group 3, ομάδα 3, τώρα είναι Chamber 3, αποφασίσαμε να έχουμε και ένα δεύτερο έλεγχο για την ε, ίδια αυτή διαδικασία. Και ακριβώς αυτά τα ευρήματα σας παρουσιάζω τώρα. Και ο έλεγχος αυτός έγινε για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η περίοδος από τη λήξη της ε, διαδικασίας, η περίοδος που είχε παρέλθει ήταν 5 με 6 χρόνια και γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι πια είχε μπει στο αυλάκι και ήταν κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τον έλεγχο αυτό. Ο δεύτερος λόγος ήταν η δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που ξεκίνησε φέτος. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο έγινε ο δεύτερος έλεγχος στη διαδικασία αυτή ήταν ότι 80% περίπου του ποσού που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περνάει μέσα από το σύστημα διαχείρισης. Δηλαδή ότι η Επιτροπή κάπου 8,5 με 9 εκατομμύρια ευρώ δαπανά το χρόνο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά πολύ ο μηχανισμός ο οποίος προσφέρει περισσότερη βοήθεια ανά τον κόσμο. 80% των ποσών αυτών όμως ε, τυχαίνουν διαχείρισης μέσω του συστήματος αυτού διαχείρισης της Επιτροπής. Ο έλεγχος έγινε λοιπόν για τους τρεις αυτούς λόγους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κίνησε γιατί, γιατί η Επιτροπή ήθελε να αυξήσει την ταχύτητα με την οποία δίνεται η βοήθεια, ήθελε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα της ε, αρρωγής και να βελτιώσει και τις δημοσιονομικές διαδικασίες. Όταν λοιπόν κοιτάμε για ποιο λόγο έγινε ο έλεγχος, ε, σας είπα ποιοι ήταν και ο στόχος μας ήταν να ε, πετύχουμε αυτά τα τρία. World Business, ταχύτητα και ποιότητα της βοήθειας. Στρέφομαι τώρα στα ευρήματα του ελέγχου. Για δύο κατηγορίες. Πρώτον, τι πέτυχε η Επιτροπή και δεύτερον, τι μένει ακόμα να γίνει. Τι έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όσον αφορά την ε, ταχύτητα, τις διαδικασίες και την ποιότητα. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν από αυτού. Όσον αφορά την ταχύτητα, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τη διαδικασία αυτή μπόρεσε να δεσμευτεί και να πληρώσει περισσότερα από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Και δίχως άλλο θα θυμόσαστε κι εσείς ότι παλιότερα υπήρχαν πολλά εμπόδια όσον αφορά την ε, απόδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα λοιπόν όλα αυτά έχουν βελτιωθεί πολύ. Δεν υπάρχουν πια αυτού του είδους τα εμπόδια. Όσον αφορά συνεπώς την ταχύτητα μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταφέρει να πληρώνει πολύ περισσότερα από ό,τι πριν ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Συνεπώς βελτιώθηκε η ταχύτητα με την οποία παραδίδεται η βοήθεια. Δεύτερον, αν δούμε τώρα τις ε, διάφορες ε, άλλες δημοσιονομικές διαδικασίες, αυτές έχουν επίσης βελτιωθεί. Όσον αφορά τώρα το τρίτο σημείο, που είναι η ποιότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, η εικόνα είναι λιγότερο σαφής από ό,τι για τα άλλα δύο σημεία. Βρήκαμε κάποιες ενδείξεις που λένε ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα, αλλά όπως θα διαβάσετε και στο έγγραφο, στον, ε, στα βρήματα δηλαδή του ελέγχου, ο τρόπος με τον οποίο ε, μετρούμε την ποιότητα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί ακόμα. Πιστεύουμε ότι βασιζόμαστε πολύ μέχρι τώρα τα εξωτερικά συστήματα διαχείρισης. Ονομάζουμε ROM. Συνεπώς, μια που έχουμε πολλές αντιπροσωπείς, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα έπρεπε και, και θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα από τις δικές μας αντιπροσωπείες. Δύο συστάσεις γίνονται. Πρώτον, οι ίδιες αντιπροσωπείες πρέπει να προχωρούν σε αξιολόγηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα όλων των παρεμβάσεων βοήθειας, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων παρεμβάσεων και να μπορεί να έρθει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα εξηγήσει και ότι η ε, κατόπιν αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της ποιότητας. Η ποιότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με, μετρήσιμους, με μετρήσιμα βέβαια στοιχεία, για παράδειγμα αναλφαβητισμός. Είναι σημαντικό να μπορούμε να μετρήσουμε τον ε, βαθμό αναλφαβητισμού. Όχι μόνο πόσα χρήματα δώσαμε, για να καταπολεμήσουμε τον αναλφαβητισμό, αλλά και πώς ο αναλφαβητισμός μειώθηκε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Έρχομαι στο δεύτερο τώρα. Τι μένει να γίνει, τι πρέπει να γίνει ακόμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ενισχυθεί. Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχουν τρεις τομείς που θα έπρεπε να προσέξουν ακόμα περισσότερο και από πλευρά τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Ένα σημείο που θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο είναι τα θέματα ελέγχου και πληροφόρησης ενημέρωσης στη συνέχεια στην Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τη στήριξη από την ε, έδρα της Επιτροπής. Και μετά υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια, που είναι μια μεγάλη πρόκληση κι αυτή. Αν δούμε λοιπόν το θέμα της διαχείρισης και της αξιολόγησης, ε, πρέπει να γίνεται συστηματικά σε επίπεδο αντιπροσωπιών. Συστηματικά, το υπογραμμίζω, όχι που και που, και με συγκεκριμένη στρατηγική για κάθε αντιπροσωπεία από τις 130-111 που είχαμε πριν. Επίσης πιστεύουμε ότι το σύστημα εσωτερικής ενημέρωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρεμβάσεις και ποσοτικά, δηλαδή με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι αυτό δεν κάνει πιο εύκολη τη ζωή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά πιστεύουμε συγχρόνω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ποσοτική έκφραση τη παρέμβαση με αποτελέσματα ποσοτικά εκφρασμένα. Να ξέρουμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Ο ρόλος στήριξης τώρα της Επιτροπής. Σελίδα 31 λέει ο μιλητής του εγγράφου μας. Πρέπει εδώ να πούμε ότι στο προσωπικό της ΔΕΦΚΟ, όπως ονομάζεται, υπάρχει υψηλό ποσοστό ε, παρουσίας του προσωπικού. με αποτέλεσμα να χρειάζεται βελτίωση όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τον πολιτικό διάλογο. Ξέρετε ότι πολλή βοήθεια είναι βέβαια οικονομική, αλλά ο πολιτικός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός γι' αυτό. Αν κάποια στιγμή αλλάξουν τα πράγματα σε επίπεδο αντιπροσωπείας όσον αφορά την ε, διαχείριση και πάμε από προγράμματα στον πολιτικό διάλογο, τότε χρειάζονται και άλλα προσόντα στο προσωπικό. Άρα οι αντιπροσωπείες πρέπει να το εξετάζουν αυτό. Και υπάρχει και το θέμα των ανθρωπίνων πόρων. Ανθρώπινοι πόροι λοιπόν, όχι ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινοι πόροι, συγγνώμη. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανθρώπινη πόροι είναι κάτι που πρέπει να περνάει από διαχείριση στις αντιπροσωπείες και υπάρχει περιθώριο ανάλυσης όσον αφορά το πώς χρησιμοποιείται το προσωπικό. Χρειάζεται και στενή συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μια μεριά και με τα κράτη-μέλη από την άλλη. Δηλαδή, η ίδια δουλειά δεν πρέπει να γίνεται και από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Κάποια κράτη-μέλη, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να κάνουν αυτά που κάνει η Επιτροπή, ούτε και η Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη. Να ανταλλάσσουν δηλαδή εμπειρίες. Άρα, μένει ακόμα εδώ να γίνει πολλή δουλειά όσον αφορά την συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Για τους ανθρώπινους πόρους, θέλω να επενθυμίσω κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση. Αν δείτε για τις αντιπροσωπείες, θα δείτε ότι 20% του προσωπικού είναι ήταν στην προηγούμενη επίπεδα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 30% ήταν συμβαλόμενοι και 50% ήταν τοπικό προσωπικό. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αν έχετε πολύ τοπικό προσωπικό, είναι προσωρινό και σε επίπεδο τη έδρας, γιατί είναι για τρία χρόνια και μετά πρέπει να φύγουν από την Κομισιόν. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνεται την εμπειρία τους, χάνεται ε, πολλή πληροφορία. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης, ότι σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την αποκέντρωση. Θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, με μερικές τελικές μου παρατηρήσεις. Από την αρχή της χρονιάς αυτής, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να εξαταστούν κάποια ζητήματα. Σε επίπεδο αντιπροσωπιών πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην διπλωματική πτυχή και στην ε, εφαρμογή. Δηλαδή στις αντιπροσωπίες αλλάζει ο ρόλος τους. Δεν ε, ε, επιδίδουν απλώς την βοήθεια μέσω προγραμμάτων σχεδίων κλπ. αναλαμβάνουν και ένα πιο πολιτικό ρόλο στο εμπόριο, με πολιτική συζήτηση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Άρα ε, ο πολιτικός ρόλος τους έχει ενισχυθεί και άρα η εφαρμογή της ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει και της βοήθειας γενικότερα παραμένει κάτι πολύ σημαντικό. και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κοιτάξουμε είναι πώς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ξεκίνησε. Πώς δηλαδή προσλήφθηκαν, ε, και θα τελειώσω με αυτό κυρία Πρόεδρε, ίσως να μην υπάρχει αρκετή εξοικείωση με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δούμε τις αντιπροσωπείες και αν δούμε τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Συνεπώς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι χρειάζεται μερικές φορές χρόνος ακόμα και για ευρωβουλευτές, ακόμα και για αξιωματούχους της ε, Επιτροπής για να μάθουν πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν προσλάβει καινούριου επικεφαλεί αντιπροσωπιών και του καταρτήσει για δύο-τρει εβδομάδε, μπορεί, λέω μπορεί, να μην φτάνει. Ακόμα και αν μπορούν να μάθουν πολύ γρήγορα. Και τέλος, τέλος κύριε Πρόεδρε, Υπάρχει και σύγχυση μερικές φορές όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της ΔΕΦΚΟ. Το συζητήσαμε με την κυρία Άστον και με τον επίδοπο τον κύριο Πίβελξ. Οπότε, η κατακλείδη δεν το έχουμε σχεδιάσει ακόμα, αλλά προβλέπουμε έλεγχο όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και για να ξανάρθω εκεί που ξεκίνησα, πρέπει να πετύχουμε την σωστή ισορροπία. Πότε έχουμε έλεγχο, τώρα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια ή αφότου έχει λειτουργήσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ήδη τρία-τέσσερα χρόνια για να έχει μπει σε μια ρουτίνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την υπομονή σας και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας για την υπομονή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρίξεν για την παρουσίασή σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα θα ανοίξω τη συζήτηση και δίνω το λόγο στην κύριο Πρέντα. Ναι, ε, είμαι ε, από το ΕΛΚΣ και ο και η συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα σήμερα σχετικά με αυτή την γνωμοδότηση του κυρίου Μαυρονικόλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ τον κύριο Πίνξεν για αυτήν την παρουσίαση που ήταν και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε μαζί μέσα στην Επιτροπή μας πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας φέτος μετά το τέλος της διαδικασίας αποκέντρωσης. Είχαμε μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο τέλος του μήνος Μαρτίου που χαιρετήσαμε με μερικές θετικές απόψεις και μερικά προβληματικά σημεία αυτής ε, της ε, μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Μετά τα όσα είπε ο συνάδελφος Μαυρονικόλας, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις ε, που θα αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών. Σχετικά με την πρώτη παράγραφο θα ήθελα να τονίσω ότι ένας από τους στόχους της ε, διαδικασίας αποκέντρωσης ε, ήταν ε, η αύξηση του αντικτύπου και της γνωστοποίησης προς τα έξω της εξωτερικής δράσης και θα πρέπει να επιμείνουμε πάνω στο σημείο αυτό κυρίως στα πλαίσια ε, της περίοδου μετά τη Λισαβόνα. Όπως τόνισε το ελεγκτικό συνέδριο, θα πρέπει να καταβάλουμε συμπληρωματικές προσπάθειες στην Επιτροπή για να αξιολογήσουμε συγκεκριμένα τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Παρέμβασης. Αυτό θα μεταφραστεί με σημαντικότερες ευθύνες όσον αφορά στην βοήθεια που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με μια μεγαλύτερη ορατότητα προς τα έξω και συμφωνώ με τα συμπεράσματα της παραγράφου 2 της γνωμοδότησης του κυρίου Μαυρονικόλα, αλλά Έχω ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας αμέσα στο πλαίσιο αυτό, διότι αυτή η γνωμοδότηση αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης στο σύνολό της και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια σύγχυση. Δεν βρίσκω ότι θα πρέπει εδώ στη δεύτερη παράγραφο να αναφερθεί το θέμα αυτό. Σχετικά με την τρίτη παράγραφο, κάθε ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρεται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, μπορεί να περιληφθεί, αλλά θα πρέπει ίσως να διαφοροποιήσουμε, να διευκρινίσουμε αυτόν τον ισχυρισμό ότι η δήλωση είναι αδύνατο απριόρι και με απόλυτο τρόπο να προσδιορίσουμε ε, ποια είναι η ισορροπία που πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στις θέσεις που αναφέρονται ε, στις πολιτικές, εμπορικές ε, θέσεις και στις αναψυξικές θέσεις. Εξαρτάται από το πλαίσιο και νομίζω ότι απαιτείται μια κάποια ευελιξία. Είναι ουσιαστικό να έχουμε μια ισορροπία που να μην προσδιορίζεται με αφηρημένο τρόπο, αλλά ανάλογα με το πλαίσιο, με το περιεχόμενο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την συνεκτικότητα της εξωτερικής πολιτικής μετά τη Λισαβόνα. Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και για να κλείσω θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο που δεν περιλαμβάνεται στη γνωμοδότηση, παρόλα τα αυτά ενέχει σημασία, θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών στις χώρες όπου υπάρχει επίσης μια πρεσβεία των ε, κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις δύο αυτές αντιπροσωπίες. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε αποτελεσματική εξωτερική αντιπροσώπευση και εξωτερική πολιτική που να είναι πράγματι συνεκτική. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λουκ Βαγκλουκ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Σημερίζεται η Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Η έκθεση αυτή δείχνει με αιτιολογημένο τρόπο ότι η αποκέντρωση από τις Βρυξέλλες προς τις αντιπροσωπείες της Ένωσης είναι μια επιτυχία. Αναφέρει ε, δικαίως ορισμένα προβλήματα η έκθεση, περιορισμένα προβλήματα μεταξύ αυτών η θέση του προσωπικού που ασχολείται με την ανάπτυξη των προγραμμάτων και αυτό αναφέρεται και από τον εισηγητή σας, τον κύριο Μαυρονικόλα, στην εισήγησή του. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι η γνώση, η εμπειρογνωμοσύνη δεν είναι πάντοτε διαθέσιμη και το turnover επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω των δημοσιονομικών ε, προοπτικών και οικονομικών είναι πιθανόν στο μέλλον η Κομισιόν να έχει πρόσθετο προσωπικό και θα πρέπει να κάνει περισσότερα και καλύτερα πράγματα με λιγότερο προσωπικό. Η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με τρεις, υπό τρεις όρους, ε, δηλαδή το προσωπικό των αντιπροσωπιών για τις αναπτυξιακές πολιτικές να χρησιμοποιούνται με καλύτερο τρόπο για τον προσδιορισμό και υλοποίηση των προγραμμάτων βοήθειας. Θα πρέπει επίσης η άσκηση Τη της Κομισιόν για καλύτερη κατανομή του προσωπικού στις αντιπροσωπίες ανάλογα με το φόρτο εργασίας των ε, διαφόρων αντιπροσωπιών να ολοκληρωθεί αυτή ε, η εργασία και θα πρέπει οι νέοι προσανατολισμοί της αναπτυξιακής πολιτικής για να αυξηθεί ο αντίκτυπος των προγραμμάτων με μεγαλύτερη συγκέντρωση ε, της βοήθειας στις χώρες εταίρους και ανάλογα με τους τομείς παρέμβασης που θα έχουν τις καλές επιπτώσει στις διάφορε αντιπροσωπείε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξαναδίνω τον λόγο στον κύριο Μαύρο Νικόλα για τα συμπεράσματα αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Ναι, νομίζω είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σίγουρα θα ήθελα καταρχήν να συμφωνήσω με όσα έχουν υποθήκη από τον κύριο Πίξτεν και η παρουσία του εδώ υπήρξε και πάρα πολύ καλά ενημερωτική, αλλά και πολύ περισσότερο μας δίνει το δικαίωμα ανταλλαγής απόψεων σε τομείς που δεν είχαμε μέχρι τώρα στην Επιτροπή την ευκαιρία να συζητήσουμε. Τώρα σε σχέση με τις κάποιες προτάσεις που ακούστηκαν από τον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος θα έλεγα ότι είναι αποδεκτές, ιδιαίτερα το θέμα που ανάφερε για τη γνωστοποίηση της εξωτερικής βοήθειας που δίνεται για το θέμα που ανέφερε για τη συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών και των διαφόρων πρεσβειών σε κάθε χώρα όπου συνυπάρχουν και όπως επίσης η προσπάθεια για να δημιουργήσουμε στο τέλος της ημέρας ένα κείμενο το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Θα περιμένουμε και τις τροπολογίες και σε κατηδία συζητήσεις για να διευκρινίσουμε οποιαδήποτε θέματα της γνωμοδότησης που κατά την κρίση κάποιων μπορεί να χρήζουν μιας βελτίωσης. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν πάρει τον λόγο μέσα από την αίσθηση ότι η δική μας δουλειά θα είναι αντιπροσωπευτική, θα είναι συνενετική για έναν τομέα που όπως ορθά ανάφερε ο κύριος Πίξτεν ε, είναι πολύ σημαντικός για την καλύτερη λειτουργία και παρουσία της δουλειάς που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα κατατεθούν οι τροπολογίε μέχρι τι 10 ε, Ιανουαρίου 2012 στι 12 και η ψηφοφορία θα λάβει ε, χώρα στις 31 ε, Ιανουαρίου και στην Επιτροπή ανάπτυξη 29 Φεβρουαρίου. Τώρα σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 11 έκθεση σχετικά με την ενδέκατη ε, δια, ε, ε, κοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παλαιστίνης που έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Νομοθετικό Συμβούλιο της Παλαιστίνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το ότι μου προσέφεραν την ευκαιρία να ε, συντάξω αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικό οι αντιπροσωπείς να καταθέτουν εκθέσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Να μην ε, υπάρχει άγνοια για τη δουλειά που γίνεται. Ε, η επίσκεψη λοιπόν περιορίστηκε στη Γάζα. Στις αρχές του έτους είχαμε επισκεφτεί τη Δυτική Όχθη. Υπάρχουν περιορισμοί ταξιδιού, δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να ε, επισκεφτεί κανείς τη Δυτική, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ ε, και την Παλαιστίνη όλα μαζί. Αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό λοιπόν ε, κάναμε δύο ταξίδια. Πήγαμε στη Γάζα, νομίζω ήταν Παρασκευή ε, Πέμπτη και Παρασκευή Νοεμβρίου, 3 και 4 περίπου. Ο στόχος ήταν να συναντηθούμε με μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, του PLC. Για πρώτη φορά λοιπόν στη Γάζα, κατά την επίσκεψή μας στη Γάζα, ε, συναντηθήκαμε με όλα τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν εκεί. Ε, σε παλαιότερες συναντήσεις συναντηθήκαμε μόνο με το Change of Reform, ήταν το όνομα της Χαμάς με το οποίο συμμετείχε στις εκλογές. Αλλά σε αυτή την ευκαιρία, σε αυτό το αξίδι που σας είπα, επιμείναμε, επειδή υπογράφηκε συμφωνία συμφιλίους μεταξύ Φατάχ και Χαμάς, τελήσαμε να συναντηθούμε ε, με όλες τις πολιτικές ε, εκπροσωπήσεις. Έτσι λοιπόν ήταν μια ιστορική συνάντηση συναντηθήκαμε με όλους ε, τους εκπροσώπους της Φατάχ, της Χαμάς, της PLP ε, και ε, με πολλούς ανεξάρτητους. Επίσης υπήρχαν και πολύ σημαντικές και ζωντανές συζητήσεις για μια σειρά θεμάτων. Εμείς λοιπόν ήμασταν βέβαια ευγενικοί ανάμεσά μας, αλλά καταστήσαμε σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει η δημοκρατία, τον πλουραλισμό την ε, ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα και την ανοιχτή κοινωνία. Μερικά από τα μέλη μας έφτιαξαν το θέμα της θανατικής ποινής και οι εκπρόσωποι της ΦΑΤΑΧ μας διαβεβαίωσαν ότι έχουν υπογράψει την ε, συνεργασία για την Ευρώπη, το Partnership for ε, Democracy, αυτό το εργαλείο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου προβλέπεται η κατάργηση της θανατικής ποινής. Άρα έχουν αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Οι άνθρωποι της Χαμάς ήταν πολύ πιο αμφίσιμοι ως προς το θέμα αυτό. Ε, τελικά ε, κάπως προέκυψε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ε, τη θανατική ποινή. Αλλά εγώ τους είπα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύει σε αυτό τα συντάγματα ή καταστατικά του το θέμα της θανατικής ποινής. Άρα δηλαδή εδώ είχαμε διάσταση απόψεων. Ένα άλλο θέμα που προέκυψε ήταν ο αποκλεισμό της Γάζας. Επίσης εξετάσαμε το θέμα της ελευθερίας λόγου, ε, των μέσων ενημέρωσης και άλλων οργανισμών. Αρκετοί, κυρίως οι ανεξάρτητοι, το κόμμα των ανεξαρτήτων και το PFLP, μας είπαν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν απόλυτα ελεύθερα στη Γάζα και χρειάζονται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Είπαν βέβαια ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να δουλέψουν ανοιχτά ε, πολιτικά αν δεν υπήρχε ο αποκλεισμό της Γάζας αν δηλαδή δεν ήταν στο έλεος των ε, μεγάλων ομάδων που ελέγχουν την περιοχή. Επίσης κατέστησαν σαφές ότι είναι υπέρ της ε, διατήρησης της αντίστασης και τους πιέσαμε, τους είπαμε τι εννοείτε, με ποιο τρόπο προτίθεστε να διατηρήσετε την αντίσταση. Αρκετοί μεμονωμένοι άνθρωποι μας είπαν ότι κατά την άποψή τους ε, υπάρχουν ανοιχτές όλες τις δυνατότητες, αλλά οι περισσότεροι επέμειναν ότι πρόκειται για ειρηνική πολιτική αντίσταση. Και όλες οι πολιτικές ομάδες ε, που ήταν παρούσες στήριξαν την πρωτοβουλία του ΑΜΑΣ στα Ηνωμένα Έθνη. Είπαν ότι 70% των Παλαιστινίων τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη πιστεύουν ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο σωστός δρόμος για να υπάρξει πρόοδος και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ε, πρέπει να πω ότι ε, εντυπωσιάστηκαν από αυτή την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών ε, να μην ε, χορηγείται πλέον ε, βοήθεια στο Παλαιστινιακό κράτος, μια απόφαση που λήφθη από την UNESCO και επικράτησε η άποψη ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αρκετά μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου είπαν ότι η Αραβική Άνοιξη δεν υπάρχει μόνο σε μία χώρα. Αυτό ισχύει κυρίως για την Ευρώπη και είπαν ότι δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στη δέσμευση στη, στην ε, υποχρέωση που έχει αναλάβει αν θέλετε η Ευρώπη απέναντι στους Παλαιστινίους. Πρέπει να τους στηρίξουμε και τους Παλαιστίνιους όπως ε, έχουμε υποστηρίξει και τους Αιγύπτιους, τους Σύριους, τους Λίβιους και άλλους. Αυτός λοιπόν ήταν ο βασικός στόχος της ε, συνάντησής μας. Είχαμε συζητήσεις ε, και με τον φορέα των προσφύγων, την UNRWA. Είπαν ότι θα διατηρήσουν το πρόγραμμα των σχολείων. Επίσης ε, είπαν ότι πρόκειται να διατηρήσουν και το πρόγραμμα υγείας. Ε, ελπίζουν μέχρι το τέλος του έτους να μπορέσουν να αποκτήσουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση γιατί αλλιώ θα αναγκαστούν να διακόψουν αυτό το πρόγραμμα. Προσφέρουν σχολική μόρφωση τουλάχιστον στα μισά παιδιά ε, σε αυτή την περιοχή. Επίσης ε, προσφέρουν εκπαίδευση στα παιδιά αυτά για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους ε, διδάσκουν για το ολοκαύτωμα, για, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και επίσης επισήμαναν ότι περίπου 10.000 παιδιά στη Γάζα δεν εντάσσονται στο σχολικό σύστημα διότι ζουν σε αυτά που αποκάλεσαν απομακρυσμένες περιοχές της Γάζας και εκεί δεν έχει πρόσβαση η ΟΝΡΑ λόγω της πολιτικής κατάστασης και διαφόρων άλλων δυσκολιών ε, που ε, μαστίζουν τους πολίτες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι η Γάζα εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή φυλακή. Δεν υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα στη Γάζα. Περίπου το 5% της οικονομικής δραστηριότητας ε, είναι μόνο το 5% αυτών που υπήρχε πριν από τον αποκλεισμό. Ε, από το Ισραήλ προς την Γάζα Υπάρχει κάποια μετακίνηση, αλλά ε, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των αγαθών που ε, χρειάζονται στη Γάζα και εισέρχονται εκεί. Βεβαίως και δεν υπάρχουν εξαγωγές από τη Γάζα και εκτός από τη βοήθεια ούτε και εισαγωγές υπάρχουν. Η Ούνρα κατόρθωσε να εισάγει κάποιο υλικό για τα κτίρια της, ε, θέλουν, προγραμματίζουν να κατασκευάσουν 100 περίπου σχολεία ε, και δεν μπορούν να τα κατασκευάσουν διότι δεν υπάρχει το απαραίτητο δομικό υλικό. Ένα σημαντικό ε, κομμάτι του υλικού αυτού προέρχεται, έρχεται μέσα από τις σύραγγες και από τα σύνορα, σύνορα με την Αίγυπτο. Όμως η ούρα δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό το υλικό γιατί είναι παράνομο. Είναι παράνομη εισαγωγή δομικού υλικού. Ε, υπάρχουν ε, περίπου 1.200 ε, σύραγγες αυτή τη στιγμή που εξακολουθούν να λειτουργούν και κατά, σε τακτά χρονικά διαστήματα οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν, επιτίθενται σε αυτές τις ε, σύραγγες αλλά ε, δεν υπάρχει κανένας άλλος ε, ε, περιορισμός. Αν είσαι στη Γάζα, εξαρτάσαι πλήρως από την βοήθεια. Δεν υπάρχει εργασία. Περίπου το 50% των πολιτών είναι κάτω της ηλικίας των 50 ετών. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της Γάζας κατ' ουσίαν καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό και τους πολίτες. Ένα από τα χειρότερα πράγματα που είδαμε είναι ότι από το Μάρτιο του 2010 29 παιδιά δολοφονήθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα διότι τα παιδιά αυτά πλησίασαν πάρα πολύ κοντά στα σύνορα. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν μια ζώνη 300 μέτρων ε, μέσα στην ίδια τη Γάζα, όχι στα δικά τους τα σύνορα, στην, στο έδαφος της Γάζας. Θεωρητικά, αν κάποιο μετακινηθεί μέσα σε αυτά τα 300 μέτρα, σε αυτή τη ζώνη, τότε κινδυνεύει να δεχθεί πυροβολισμούς. Και υπάρχουν ε, πανό που το λένε. 19 πάντως από τα 29 αυτά παιδιά, 13 με 17 ετών, ήταν εκτός της ζώνης αυτής, στα 600 μέτρα από τα σύνορα. Τα παιδιά αυτά πυροβολήθηκαν στα χέρια, στα πόδια, κάποιο μάλιστα δέχτηκε πυροσβολισμό στο κεφάλι. Κανένα ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή του, αλλά καταλαβαίνετε τι τραύμα είναι αυτό για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους που έπρεπε να τα φροντίσουν μετά. Συνεπώς, πρέπει να πω πριν ολοκληρώσω και από εκεί και πέρα ευχαρίστω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με ομάδες γυναικών. Πήγαμε σε ένα από τα σχολεία της, πήγαμε και είδαμε και έργα που γίνονται για τα ύδατα στην Κάζα. Πρέπει να ξέρετε ότι η υδραγωγή είναι κατεστραμμένη και ότι αν πολύ γρήγορα δεν γίνει κάτι, τότε θα μολυνθεί το νερό. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερή η κατάσταση στη Γάζα. Δεν ξέρω τι λύση άλλη μπορεί να υπάρχει πέρα από τη διεθνή κοινότητα να ζητήσει να σταματήσει ο αποκλεισμός αυτός. Ο Σαλή επέστρεψε στην οικογένειά του ευτυχώς και από εκεί και πέρα η διεθνής κοινότητα μπορεί να πει ότι πρέπει να σοβαρευτούμε με την κατάσταση στη Γάζα και ο κόσμος εκεί να μην τυχαίνει της μεταχείρισης που τυχαίνει τώρα. Και κάτι τελευταίο που θα πρέπει να σας πω είναι το εξή. Συναντηθήκαμε και με κάποιους από τους κρατούμενους που μόλις απελευθερήθηκαν από τις φυλακές μετά την ανταλλαγή που έγινε για τον Σαλίτ ήταν από πολύ νέους μέχρι λιγότερο νέους. Κάποιος μάλιστα είχε περάσει 20-25 χρόνια στη φυλακή. Ήταν ε, μια όντως ε, έτσι, σύντομη συνάντηση. Είπαν πώς αποφασισμένοι είναι για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Ορισμένοι ήταν και πολύ θυμωμένοι επειδή δεν ε, δίνουμε αρκετή προσοχή ε, στο θέμα των κρατούμενων, κάπου 5.000 είναι στις Ισραηλινές ε, φυλακές και κάπου 150 είναι παιδιά. 22 άτομα δε είναι εκλεγμένοι. Έχουν όμως συλληφθεί τότε όταν για να, ως αντίδραση στην κράτηση του Σαλίντ. Ίσως η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να μπορούσε να ξεκινήσει μια έκθεση. Γιατί εκείνοι δεν μπορούν. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ίσως η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων λοιπόν να μπορεί να ξεκινήσει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την κατάσταση στη Γάζα. Φαντάζομαι ότι θα θέλουν πολύ να το στηρίξουν αυτό και να βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας τέτοιας έκθεσης. Πάντως πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά γιατί η κατάσταση εκεί είναι πολύ άσχημη και δημιουργεί μια νέα γενιά νέων που μεγαλώνουν μέσα στο μίσος για το Ισραήλ. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση γρήγορα, εκεί θα καταλήξουμε. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε δύο κράτη, το Ισραήλ που να μπορεί να ζει ειρηνικά με την Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση μακροπρόθεσμα. Ούτε μπορούμε τώρα ε, να κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να σταματήσει αυτή η κατάσταση ε, στη Γάζα. Ευχαριστώ για αυτήν την έκθεση. Δίνω τον λόγο στην κυρία Κλίνικρε. Με συγχωρείτε. Ναι, ήθελα να προσθέσω μερικά στοιχεία εφόσον κατά την ίδια περίοδο η Επιτροπή ε, ε, δικαιωμάτων της γυναίκας και ισότητας των φίλων ε, των, της οποίας είμαι μέλος επισκέφθηκε την Γάζα, την Δυτική Όχθη εφόσον η Επιτροπή Γυναικών ήθελε να ενημερωθεί για την κατάσταση των γυναικών στην ε, περιοχή αυτή και τα προβλήματα των γυναικών. Γι' αυτό υποφελούμε για να προσθέσω σύντομα μερικές πληροφορίες σχετικά με τις γυναίκες στη Γάζα, εφόσον συναντήσαμε την Επιτροπή Γυναικών της Γάζας και συναντήσαμε και επισκεφτήκαμε μάλλον έναν ε, χώρο που η Ούνρα εργάζεται για τις ε, γυναίκες, ε, για την χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φίλων και θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες στην Γάζα υφίστανται διπλή καταπίεση την καταπίεση που υφίστανται πολλές γυναίκες στον πλανήτη λόγω της πατριαρχικής οικογένειας και μια διπλή καταπίεση εφόσον υφίστανται και την καταπίεση αυτού του αποκλεισμού που είναι απάνθρωπος και η κατάσταση των γυναικών στην Γάζα δεν γίνεται πολύ λόγος για αυτήν, αλλά είναι πράγματι τρομερή. Όπως είπε και ο κύριος Ντερόσα πριν από λίγο, ε, ο μεγαλύτερο ε, ποσοστό του πληθυσμού στην Γάζα είναι παιδιά, παιδιά που πρέπει να τραφούν, να ανατραφούν, να εκπαιδευθούν και οι γυναίκες ασχολούνται με τα παιδιά και αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, κάνουν ουρές ε, για να λάβουν την επισητιστική βοήθεια της ευρωπαϊκής που παρέχει σε μεγάλο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προοπτικές, οι μελλοντικέ δεν υπάρχουν για τα παιδιά αυτά και οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ε, δυσκολίες λόγω της ανεργίας που είναι πάρα πολύ σημαντική στην Γάζα. Η κατάσταση λοιπόν των γυναικών είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα ήθελα να επιμείνω πάνω σε αυτό το σημείο. Υπάρχει επίσης και μια ιστορία που θα ήθελα να πω που θα σας εκπλήξει αν είδατε το φίλμα. Λοκοσόν το Γαζά, το γουρούνι της Γάζας ε, που προβάλλεται στην Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Για αυτούς που είδαν το έργο αυτό θα ήθελα να πω ότι το έργο αυτό που είναι κομικό έργο στην πραγματικότητα ε, το περιεχόμενο, το πλαίσιο που παρουσιάζεται στην, στο αυτή αντιποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, δεν είναι σωστή εικόνα που παρουσιάζεται. Για αυτούς που είδαν την ταινία θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια μικρή ιστορία που αναφέρεται στην αγορά ενός προϊόντος που ονομάζεται Viagra. Βλέπουμε κάπου ένα παιδί που αγοράζει Viagra στο φαρμακείο και δεν είναι κατά τύχη που ο σκηνοθέτης το έβαλε αυτό στην ταινία. Οι γυναίκες στη Γάζα μου είπαν ότι όντως το Viagra είναι ένα από τα προϊόντα που ε, διέρχεται από τις σύραγγες κάθε μέρα, διότι οι άνθρωποι, οι άντρες βαριούνται στη Γάζα, δεν έχουν τίποτα να κάνουν και οι γυναίκες δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς με την καθημερινή του ζωή ε, σε αυτήν την ε, περιοχή, σε αυτό το γκέτο που είναι η Γάζα. Αυτό είχα να προσθέσω στην έκθεση του κυρίου Ντερόσα. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους κύριε Κίνησον, τον κύριο Ντερόσα για την εισήγησή τους, για τα όσα μας είπαν. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι αλληλέγγυη με τον λαό της ε, Γάζας με τρόπο ίσως δυσανάλογο. Είναι όνειδος, όνειδος για όλους μας, αλλά θα ήθελα μάλλον να μιλήσω για έναν λαό που σέβομαι πάρα πολύ ε, και ε, που είναι ο λαός του Ισραήλ για τον οποίο έχω φιλικές διαθέσεις και δεν νομίζω ότι η κατάσταση που υπάρχει στην Γάζα τώρα δεν είναι προς όφελος του λαού του Ισραήλ. Δεν το πιστεύω αυτό. Φοβούμε επίσης ότι η κατάσταση στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής θα παραμείνει στάσιμη για πάρα πολύ καιρό εφόσον οι Αμερικανοί με τις επερχόμενες εκλογές βρίσκονται σε πλήρη παράλυση. Νομίζω ότι η κυρία Άστον ενδιαφέρεται βεβαίως, ενδιαφέρεται πραγματικά για τα όσα συμβαίνουν και θέλει να προωθηθούν τα πράγματα, η διαδικασία σχετικά με αυτήν την διαμάχη, αλλά είναι νομίζω και αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκαν να σκεφτούν out of the box λόγω των προβλημάτων που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για το Κοινοβούλιο αυτό να παίξει το ρόλο του και να αναλάβει πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι ο κύριος Ντερόσα έχει δίκιο που προτείνει αυτή ε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αναλάβει μια πρωτοβουλία ε, για μια έκθεση στην Γάζα και να ασκήσει πίεση για τα θέματα ουσίας, ούτως ώστε να ρυθμιστούν. Πιστεύω επίσης ότι εκτός από την ίδια την κατάσταση στη Γάζα, όσον αφορά και τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Πελαστίνη, υπάρχει επίσης και το θέμα της Αραβικής Άνοιξης που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είδα ένα ντοκιμοντέρ τρομερό στην BBC, στο BBC νομίζω για την κατάσταση lawlessness ε, στο Σινά, δηλαδή όπου, όπου δεν υπάρχει δίκαιο ε, και εκεί με τους εμπόρους, τους διακινητές μεταναστών που τους διακινούν για να τους κλέψουν τα οργανά τους και αυτό δείχνει τον τρομερό κίνδυνο που ελοχεύει για όλους, για τους μετανάστες αλλά και για όλους, ακόμη και για το Ισραήλ. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να εξακολουθήσουμε να κλείνουμε τα μάτια. Θα πρέπει να αναλάβουμε ε, πρωτοβουλία έκθεσης όπως ο κύριος Ντερόσα το πρότεινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Λαντμπέργκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ντερόσα, διότι είχε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να πάει στη Γάζα, να μιλήσει με πολιτικούς επιτόπου, να μιλήσει με εκπροσώπους της Χαμάς. Τώρα η Χαμάς ε, και η Φατάχ ε, έρχονται πιο κοντά, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε για το εξής. Αν έχουν και οι δύο σαφή άποψη για το εδαφικό, για τα σύνορα, πώς θα χαραχθούν τα σύνορα, έχουν την ίδια άποψη για το πώς θα συμβιώσουν με τα όμορα κράτη που θα είναι αναγνωρισμένα με ίσους όρους συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Έχουν κοινή θέση η Φατάχ και η Χαμάς. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι στη μελλοντική Παλαιστίνη θα έχουμε μία και μόνο ηγεσία και όχι δύο αντιμαχόμενες ηγεσίε με διαφορετική προσέγγιση προς το Ισραήλ γενικότερα προς τις γειτονικέ χώρες. Η Γάζα ή η Παλαιστίνη είναι έτοιμες για να γίνουν η πατρίδα εκατομμυρίων προσφύγων που ζουν τώρα σε καταπλησμούς. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την προοπτική. Και ερωτώ, αν αυτό το κράτος αντιμετωπίζει ως κράτος όπου θα πάνε όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, θα πρέπει να ε, ενσωματώσει στο έδαφος του όλα αυτά τα εκατομμύρια. Η Γάζα είναι ήδη ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη. Επικρατεί συμφόρηση στη Γάζα. Όσον αφορά τις προοπτικές ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους, ε, τη δυνατότητά του, την ικανότητά του να συνάπτει ε, διεθνείς συμβάσεις για θέματα στρατιωτικής ασφάλειας, ας πούμε, με το Ιράν ή με τη Ρωσία ή με την Κίνα. Η Παλαιστίνη θα αναλάβει την υποχρέωση στα πλαίσια της αμοιβαίας αρρωγής η μία χώρα να υπερασπίζει την άλλη. Η Παλαιστίνη θα εμφανιστεί με διεθνές πρόσωπο και θα ενταχθεί την ομπρέλα των ΟΕΕ. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό. Θα συνεπάγεται μεγαλύτερη ειρήνη ή περισσότερες απειλές στην περιοχή. Και θέλω να ρωτήσω, στις ε, συζητήσεις ε, που είχατε με τη Χαμάς, άραγε τοποθετήθηκαν ε, σε πυροβολισμούς από την άλλη πλευρά των συνόρων προς το Ισραήλ, προς παιδιά, γιατί δολοφονήθηκαν και παιδιά στο Ισραήλ με αυτούς τους ε, πυροβολισμούς που ξεκινούσαν από τη Γάζα. Αυτές λοιπόν τις πράξεις ε, τις εγκρίνουν ή τις ε, καταδικάζουν. Θα προσπαθήσουν να τις σταματήσουν. Ίσως λοιπόν είναι μια ευκαιρία για μας να μας πείτε εσείς άμεσα που επισκεφθήκατε την περιοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ κύριε Λαντμπέργκς. Μήπως ο κύριος Ντερόσα θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, πολλά σημεία σχετικά το LFC, ε, η Χαμάς, ε, η Φατάχα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Ε, μιλάω για όλες τις πολιτικές ομάδες ανεξάρτητων πεπιθήσεων που είναι εκλεγμένες, όχι μη εκλεγμένες οργανώσεις που επιδίδονται στη βία. Θα ήθελα να διευκρινίσω ε, το θέμα εδώ ως ε, ε, Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι δυνατόν για μας να οργανώσουμε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση με εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων της Δυτικής Όχθης, της Γάζα, εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν εφικτό αυτό να γίνει το 2006 εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήταν μια άσκηση πάρα πολύ χρήσιμη να έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ και θα μπορούσατε να θέσετε τις ερωτήσεις αυτές ε, στα άτομα αυτά και όχι σε μένα που είμαι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι εγώ σας λέω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλων οργανώσεων για τις οποίες δεν έχω ευθύνη. Θα σας στείλω βεβαίως ένα αντίγραφο της έκθεσης, της συνάντησης που είχαμε, όπου απόψεις, διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν από διαφορετικές οργανώσεις. Και Βεβαίω, όποιο μέλο θέλει αυτή αυτό, το αντίγραφο μπορεί να μου στείλει ένα email και θα σα στείλω το αντίγραφο αυτό και σε πολλά μέλη. Επίση, το θέμα είναι ότι διευκρινίσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αντίθετο προς την βία ε, στην αναζήτηση του Παλαιστινιακού κράτους. Πάρα πολλά μέλη, ακόμα και μέλη της Χαμάς, του PFLP και της Φατάχα, είπαν ότι ήταν υπέρ της ειρηνικής αντίστασης στην κατοχή, υπέρ των διαπραγματεύσεων. Ε, υπήρξαν διάφοροι βαθμοί απόψεων που εκφράστηκαν σε σχέση ε, με την δέσμευση όσο προς τα σύνορα του 67 ενός κράτους μέσα στα σύνορα του 67. Η Χαμάς είναι κάπως πιο ασαφής αλλά πάντως έχουν κάνει ε, δηλώσεις στην ηγεσία τους ότι θα δεχόντουσαν ένα Παλαιστινιακό κράτος ε, με βάση τα σύνορα του 67. Υπήρξαν βεβαίως διχογνωμίες ε, σε σχέση με το τι είναι αυτή η δέσμευση και το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα πράγματα με βάση αυτό το θέμα σε σχέση με τις σχέσεις της Γάζας με το Ισραήλ και ότι πρέπει το διεθνές δίκαιο να τηρείται από όλου ε, σε μια ρύθμιση ε, του, ε, του, και θα πρέπει και το Ισραήλ να σέβεται το διεθνές δίκαιο και ότι δεν θα πρέπει οι άμαχοι να κινδυνεύουν. Θα πρέπει δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία επίθεση από την Γάζα στο Ισραήλ. Εμείς ως εκπρόσωποι αυτού του Κοινοβουλίου νομίζω παίξαμε το ρόλο μας διότι διαβιβάσαμε τη στάση, την άποψη αυτού του Κοινοβουλίου και διευκρινίσαμε ότι ο πληθυσμός της Γάζας όσον αφορά αυτό το κοινοβούλιο. Εμείς ασχολούμεθα με τον, τον λαό της Παλαιστίνης. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζουμε τη μία ομάδα ή την άλλη αλλά την Παλαιστίνη αυτή καθεαυτή και τον πληθυσμό της Παλαιστίνης. Και να πω και στους ίδιους τους Παλαιστίνιους τι μέλλον, πολιτικό μέλλον θέλουν. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να περιμένουμε μια κοινωνία να είναι ενοποιημένη, ενωμένη πολιτικά. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία στην Ευρώπη, η κοινωνία στην Ευρώπη που να έχει ένα μόνο πολιτικό κόμμα. Έχουμε όλοι δωδεκάδες πολιτικά κόμματα που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο και είναι η κατάσταση στο Ισραήλ και θα πρέπει να είναι και η κατάσταση στην Παλαιστίνη με 14 διαφορετικές πολιτικές ομάδες στη Δυτική Όχθη, στην Γάζα και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το να προτείνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική δύναμη, ε, ότι όλοι να ενωθούν κάτω από την αιγίδα της Φατάχ, αυτό δεν είναι ρεολιστικό. Αλλά με την συμφωνία συμφιλίωσης θα πρέπει να συμφωνήσουν για τα πολιτικά περαιτέρω βήματα για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Υπάρχει ανάμεσα στην Χαμάς, στον Χάνιε, για να συζητήσουν ε, ε, τον μηχανισμό για εκλογές, διευθέτηση για μια εκλογική επιτροπή που θα παρακολουθήσει αυτές τις εκλογές και ελπίζω το κοινοβούλιο αυτό να μπορέσει να ε, στείλει ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν αυτές τις εκλογές Νομίζω ότι ένα από τα κρίσιμα θέματα θα είναι ε, όταν λάβουν χώρα αυτές οι εκλογές είναι ότι όσοι θα συμμετάσχουν θα χρειάζονται μια εξασφάλιση, μια εγγύηση από την διεθνή κοινότητα, από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα τηρηθεί, πράγμα που δεν έγινε την τελευταία φορά. Και αυτό ήταν εις βάρος μας, εις βάρος της Ευρώπης. Δεν τηρήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν έγινε σεβαστό. Δεν, δεν χρειάζεται βεβαίως να επαναλαμβάνουμε τα όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή θέση προς όφελος μιας ειρηνικής ρύθμισης στην Παλαιστίνη και εμείς θα πρέπει ε, να τηρήσουμε, να σεβαστούμε το αποτέλεσμα των επιλογών του Παλαιστινιακού λαού, ή θα παίζουμε διπλό παιχνίδι. Δεν θα ε, δεν θα, δεν θα, εμείς δεν θα σεβόμεθα την δημοκρατία όπως ζητούμε τους άλλους να τη σέβονται. Αυτό ήθελα να τονίσω και ένα τελικό σημείο. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, να έχει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ίσως δεν, εγώ δεν είμαι μέλος ε, της Επιτροπής, δεν μπορώ να επιμείνω, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλή ιδέα. Δύο μικρά σημεία πρωτού κλείσω. Ε, αυτό που αμελήσαμε να αναφέρομαι είναι ότι επισκεφθήκαμε δύο πανεπιστήμια στη Γάζα και με περίπου 50.000 ε, νέους στη Γάζα, στα πανεπιστήμια και ε, λιγότεροι ε, ε, από 10% των αποφύτων πανεπιστημίων μπορούν να βρουν δουλειά. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι κανένας φοιτητή πανεπιστήμιου στη Γάζα δεν επωφελείται από το πρόγραμμα Έρασμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ πολλές χιλιάδες από το Ισραήλ επωφελούνται. Ε, Βεβαίω, ε, εκτός από τη Γάζα, πάρα πολλοί δεν μπορούν να ταξιδέψουν ε, κάποια ηλικία και να έρθουν στα πανεπιστήμια. Ε, οι ε, ομιλητέ, οι καθηγητέ μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά οι φοιτητέ δεν μπορούν να υποφεληθούν από αυτήν την αλληλεπίδραση ε, που υπάρχει από το πρόγραμμα Έρασμό. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συζητηθεί με τι αρχέ του Ισραήλ, ούτω ώστε να μπορούν οι φοιτητέ αυτοί να ταξιδέψουν. Και τελικά τελικά, τελικά ένα θέμα το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Γάζα αλλά με το θέμα της ειρήνης και της συμφιλίωσης μεταξύ του Ισραήλ και της ε, Παλαιστίνης. Είναι το θέμα των Βεδουινών. 200.000 ε, Βεδουίνοι ε, ζουν και στο Ισραήλ και 30.000 από αυτούς σε περιοχή υπό στρατιωτικό έλεγχο Ισραηλινό στην Δυτική Όχθη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση θέλει να στείλει 30.000 από αυτούς στο Νεγκεύ, στον έρημο του Νεγκεύ σε χωριά με ανεγνωρισμένα ε, που χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς εγκαταστάσεις, ε, χωρίς ε, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, χωρίς νερό, χωρίς καν ηλεκτρισμό. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να εξεταστεί. Το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να επιμείνει για συμμόρφωση προς τους κανόνες και τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η δύναμη της Ευρώπης είναι να επιμείνει πάνω στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών κανόνων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και κάνω έκκληση από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ούτω ώστε οι Παλαιστίνοι ε, και οι Άραβες του Ισραήλ να την χάνουν ε, ίσης και δίκαιας μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάνοκ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Το έχω πει επανειλημμένα στο παρελθόν ε, την ε, δημοκρατία τη φιλελεύθερη και την πλουραστική δημοκρατία δεν τη θεωρώ απλά μια άσκηση ψήφου. Περιλαμβάνει και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίε και επίση και το σεβασμό για τα δικαιώματα των μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των ε, ομάδων, θρησκευτικών ομάδων και κυρίω ε, των δικαιωμάτων ε, των γυναικών. Γιατί Χαμά, το έχω πει, έχω προειδοποιήσει, είναι όπω η Ήρα, ήταν τρομοκρατική οργάνωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρωτήσει την ε, Χαμάς επίσης ε, τρομοκρατική οργάνωση. Δεν έχει τροποποιήσει το καταστατικό της και δεν θέλουν το εβραϊκό κράτος. Ε, στηρίζουν την αντισημιτική ιδεολογία. Γι' αυτό εγώ ή οποιοδήποτε άλλος με το δικό μου το ιστορικό και την προσωπικότητα γιατί να πρέπει να σεβαστώ αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ τουλάχιστον με το δικό μου το λεξιλόγιο αυτό δεν το λέω δημοκρατία. Στην Αίγυπτο βλέπουμε και εκεί υπάρχει μία άνοδος του Ισλαμισμού και φοβάμαι ότι αν αυτοί αναλάβουν εξουσία δεν θα έχουμε δημοκρατία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα για το τι ακριβώς είναι η δημοκρατία. Είναι μόνο οι εκλογές ή είναι τα κόμματα που δεσμεύονται για θεμελιώδεις ε, ελευθερίες. Επίσης, ε, πολλοί όταν αναλαμβάνουν εξουσία δεν φαίνουν νόμους οι συμβάσεις και γι' αυτό όταν καταλαμβάνουν εξουσία σχεδόν πια δεν μπορεί κανένας να ξεφορτωθεί πια όπως συμβαίνει στη Δύση. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Αν επανεκλεγεί λοιπόν η Χαμάς ε, φοβάμαι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα γιατί ένα μεγάλο, σκεπτικό, ένα μεγάλο κομμάτι του σκεπτικού τους είναι ξένο για μας. Μία απάντηση. Κυρία Okay να απαντήσω κι εγώ. Ε, κάποιοι ε, για τους Ισραηλινούς, κάποιους τουλάχιστον, δεν υπάρχει Παλαιστίνη στον χάρτη. Εντάξει, για μερικούς υπάρχει, αλλά γενικά δεν ε, την αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία. Και έχω και να κάνω και μια παρατήρηση για αυτά που είπε ο κύριος Λανσπέργκερ. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία άνα όσοι έρχονται από τις χώρες που βρίσκονταν υπό κατοχή επί Σοβιετικής Ένωσης ε, σκεφτείτε, να προσπαθήστε να νιώσετε λιγάκι πώς νιώθουν και αυτοί στη Γάζα που βρίσκονται ε, σε τέτοιον αποκλεισμό. Δείτε τι βία έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος των πολιτών, μα πρόκειται για κατοχή. Αυτό κάνουν. Ρουκέτες εντάξει. Τις καταδικάζουμε. Το λέμε αυτό. Αλλά μπορείτε να το δείτε κι αλλιώς. Χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό, ελικόπτερα, Ισραηλινοί. Δεν είναι καλύτερο από τις ρουκέτες που πετάνε οι Παλαιστίνοι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο λοιπόν αν ε, όσοι έρχονται από τις χώρες που βρίσκονταν υποκατοχή επί Σοβιετικής Ένωσης να δείξουν ε, λίγο κατανόηση και να νιώσουν λιγάκι πώς νιώθουν και οι άνθρωποι αυτοί στη Γάζα που βρίσκονται υποκατοχή. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το βάζαμε στο ψηφισμό μας. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό νομίζω όταν μιλήσατε κύριε Λαντμπέργκερ ήταν το θέμα των ε, καταβλισμών. Η Επιτροπή μας πρέπει να το χειριστεί αυτό. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί κανένας άλλος δεν ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσοι πολλοί, κυρίως στο Λίβανο, αλλά και αλλού. Τι τύχη τους περιμένει αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν, ναι, και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό το δικαίωμα, αλλά πώς γιατί εξαρτόμαστε από τη λύση. Εμείς τι θα τους πούμε. Θα πούμε στο Λίβανο ή θα τα αφήσετε όλα, ε, θα φύγετε από εκεί. Πώς θα γίνει. Ποιο είναι το δικό μας όραμα για τόσο πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ποιο θα είναι το μέλλον των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε δεν είναι με χρήματα που θα βοηθήσουμε, όχι. Και λυπάμαι που δεν ήμουν από την αρχή, αλλά και εγώ ήμουνα στη Γάζα από την Επιτροπή Γυναικών που επισκέφθηκε την Γάζα και την περιοχή και στηρίζω αυτά που είπε ο Πρίνσιας για τους Βεδουίνους, για παράδειγμα, και για τις γυναίκες το Ισραήλ τι λέει, εμείς δεν ανακατευόμαστε για τις γυναίκες ε, μέσα στους βιδοίνους γιατί είναι δικά τους πολιτιστικά ζητήματα. Ενώ θα έπρεπε να στηρίζει τις ε, γυναίκες αυτές, οι οποίες είναι το μέλλον των Βεδουίνων. Είναι εκπληκτικός πληθυσμός που χρειάζεται τη στήριξή μας. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους. Θα θέλω να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί Όχι, ο κύριο Ντερόσα ίσω. γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που περιμένουν για τις δικέ τους εκθέσεις. Πολύ σύντομα κύριε Ντερόσε. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομο. Θέλω να επαναλάβω. Με τίποτα δεν είμαι εγώ εκπρόσωπο της Χαμάς, ούτε και τη Φατάχ εξάλλου. Απλώς μεταφέρω τις ε, σχέσεις μας και τις ε, αξίες του Κοινοβουλίου προς το Νομοθετικό Συμβούλιο της Παλαιστίνης. Αυτό κάνω και νομίζω ότι το κάνω καλά. Θέλω επίσης να πω, κοίταξτε ο κύριος ε, και έκανε μια σύγκριση με την Ήρα. Εγώ είμαι Ιρλανδός και από το 69 που φτιάχτηκε, να ξέρετε ότι όλη μου την πολιτική ζωή την πέρασα προσπαθώντας να τους πολεμήσω. Και ναι, το 94 ήμουνα στην κυβέρνηση, μίλησα μαζί τους και διαπραγματεύτηκα την ειρήνη μαζί τους. Βλέπετε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Χαμάς είναι μια οργάνωση που θεωρεί τον εαυτό της απελευθερωτική είναι ένα μείγμα ανθρώπων που είναι από δημοκράτες σε αντιδημοκράτες. Έτσι είναι συνήθως τέτοιες οργανώσεις, οπότε πρέπει να προσπαθήσει κανείς να συνδεθεί με εκείνου από αυτούς που θέλουν μια δημοκρατική και ανεξάρτητη Παλαιστίνη και να απομονώσουμε τους υπόλοιπους. Δεν μπορείς να το κάνεις αν βάλεις την απομόνωση ολόκληρη την οργάνωση και πεις ότι δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί έχει στον τίτλο της Χαμάς. Όχι, πρέπει να βρούμε διάβλους για να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και να διαπραγματευτούμε μαζί τους μια ειρηνευτική λύση. Γιατί δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια λύση για την ίδρυση του κράτους της Παλαιστίνης με 40% να μένουν εκτός της διαπραγμάτευσης. Δεν γίνεται πρέπει να πετύχεις ευρεία συνένεση και με όλους τους Παλαιστινίους αλλά και με όλους τους Ισραηλινούς. Οπότε, παρακαλώ, μην δαιμονοποιούμε τα διάφορα στοιχεία που συμμετέχουν σε αυτή την φρικτή διένεξη είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Εμείς έχουμε ένα θετικό ρόλο να παίξουμε να φέρουμε το κόσμο μαζί να συζητήσει και να βρει λύση και όχι αντίθετα να τους απομακρύνουμε τους μένα από τους δε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Ιντερό και περνάμε στο επόμενο σημείο, σήμερα 12, που είναι η έκθεση σχετικά με την τέταρτη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίηση και Σύνδεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αλβανία, που έλαβε χώρα στα Τύρανα στι 8 και 9 Νοεμβρίου. Το λόγο έχει ο κύριο Κούκαν, ο οποίο προείδρευε τη αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι πρόσφατα η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αλβανία χαρακτηρίζεται από ένταση. Αυτό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009 με τις κοινοβουλευτικές εκλογές και μετά ε, το κόμμα της αντιπολίτευσης ε, άρχισε να μποϊκοτάρει τη δουλειά της κυβέρνησης. Κλιμακώθηκε η κατάσταση τον Ιανουάριο αυτού του έτους. Η αστυνομία δολοφόνησε διάφορους ε, κατοίκους, πολίτες, κατά διάρκεια διαδηλώσεων. Φέτος οι εκλογές του Μαΐου στην Αλβανία και πάλι κρίθηκαν ε, νοθευμένες από το σχελιστικό κόμμα της Αλβανίας. Έτσι λοιπόν η Αλβανία δεν προτάθηκε για να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας σε δύο συνεχείς εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάστηκαν στενά για να βρουν ε, κοινό έδαφος ε, ανάμεσα στις ε, δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Τους τελευταίους μήνες, χάρη σκληρής διπλωματικής δουλειάς της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ατριανά, κυρίως του πρέσβη κ. Σεκουή και χάρη της δουλειάς Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Γενικού Διευθυντή κυρίου Σανίνο, με τη βοήθεια αυτών λοιπόν επιτέχθηκε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές προχωράει η κοινοβουλευτική εργασία με τη συμμετοχή, έκτοτε με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η ΣΑΠΚ, κατόρθωσε να εκδώσει ε, κοινή δήλωση. Και αξίζει να αναφερθούμε σε αυτήν, διότι σε τρεις ε, παλαιότερες ε, περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί κοινή δήλωση λόγω των ε, ε, ασυμβίβαστων απόψεων ανάμεσα στους, ε, στις αντιμεχόμενες πλευρές Αλβανίας. Η συνάντηση λοιπόν έλαβε χώρα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου και προβλήθηκε ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης και επίσης γενικότερα. 14 εταίροι της Αλβανίας συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση. Υπήρξαν συζητήσεις με τον πρόεδρο της Αλβανίας, τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον Υπουργό Δικαιοσύνη και τον ε, αναπληρωτή Υπουργό, ε, αναπληρωτή Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας που μας δέχτηκε, ε, τον κύριο Μπερίσα, ο οποίος όταν επισκεφτήκαμε την Αλβανία έλειπε από τη χώρα. Οι βασικότερες συζητήσεις εστιάστηκαν σε θέματα που αφορούν στις ε, μεταρρυθμίσεις στο ε, κοινοβούλιο στην Αλβανία. Όλα τα μέλη ε, παρουσίασαν μια πολύ επικοδομητική στάση και μίλησαν όλοι με μία φωνή. Αυτό το εκτίμησα ιδιαίτερα και θέλω να τους ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας εδώ, τους ευρωβουλευτές. Όπως σας είπα, στο τέλος προέκυψε κοινή δήλωση και αυτό ήταν πάλι η επιβεβαίωση μιας νέας πιο θετικής πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Σε γενικές λοιπόν γραμμές ήταν μια αρκετά επιτυχημένη επίσκεψη. Και εάν η συνεργασία των δύο αντιμαχόμενων πλευρών οδηγήσει σε σταθεροποίηση του πολιτικού κλίματος στην Αλβανία, τότε η χώρα θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να κάνει ένα θετικό βήμα ε, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Και φαντάζομαι θα ήταν χρήσιμο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να εγκρίνει ένα ψήφισμα για την Αλβανία πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μια εύθραυστη συνεργασία ανάμεσα στα δύο μπλοκ. Έχουμε νέα εκλογική νομοθεσία, εκλογές προέδρου. Ε, πολλοί άνθρωποι λοιπόν, κυρίως οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στα Τύρανα, ήταν επιφυλακτικοί ε, για την βιωσιμότητα της συνεργασίας. Την έκριναν ε, επιπόλαιη, επιφανική και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ε, σε αυτό τον δρόμο η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, αν αμφισβητηθεί στην Αλβανία ο συσχετισμός δυνάμεων, εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι ε, συγκρατημένα αισιόδοξο. Και οι δύο πολιτικοί ηγέτες συνεργάζονται, χωρίς βέβαια ιδιαίτερο ενθουσιασμό, όμως, εν πάση περιπτώσει, συνεργάζονται και αποδίδουν συνεργασία τους. Άρα δηλαδή για μας, και αυτό είναι το καταληκτικό μου μήνυμα, είναι απαραίτητο όλοι οι ενωσιακοί θεσμοί συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και όλων των πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, του ΕΛΚ, όλοι πρέπει να μιλάμε με μία φωνή και να στείλουμε το ίδιο μήνυμα σε όλους τους πολιτικούς παίκτες στην Αλβανία. Και πρέπει να αποφύγουμε λάθος μηνύματα ή ατυχήματα αν θέλετε. Και αυτό για να μην βλάψουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Η χώρα έχει χάσει δύο χρόνια λόγω της ε, πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων ε, πολιτικών συνασπισμών. Φτάνει πια όμως, διότι αξίζει κάτι καλύτερο στους πολίτες της ε, Αλβανίας. Νομίζω η κατάσταση άλλαξε μετά το μήνυμα που εξέπεμψαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είδαν στα μάτια τους την πραγματικότητα και κατανόησαν ότι αν δεν υπάρξει σοβαρός πολιτικός διάλογος ανάμεσά τους, δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ε, ας ε, μην φροντίσουν μόνο να καταστρέψουν τις ελπίδες. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Τώρα το δίνω τον λόγο στον κύριο Ποστινάρου που ήταν αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω τα σχόλια του Προέδρου κ. Κούκαν και να πω ότι συμμερίζομαι πλήρως τα σχόλιά του και τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε μια ειδική συνάντηση που για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η συνάντηση με τον πρόεδρο όχι το, ο πρόεδρος, όχι πολιτικό κόμμα, ο πρόεδρος έπαιξε ένα ρόλο εξισορρόπησης για να περάσει αυτήν ε, την ε, κρίση, βαθιά ριζωμένη κρίση στην Αλβανία. Και ο πρόεδρος ε, ανέφερε τρεις απόψεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή. Πρώτα, ότι στο στιγμή κλειδί για την βιωσιμότητα της διαδικασία ανάμεσα στα δύο πολιτικά κόμματα και την υλοποίηση των 12 προτεραιοτήτων κλειδιά θα είναι η υιοθέτηση των αλλαγών για τον εκλογικό νόμο συν η εφαρμογή των απαιτουμένων υποδομών. Δηλαδή ο, ο νόμος και ο μηχανισμός που πρέπει να υπάρχει. Δεύτερον, ο πρόεδρος ανέφερε ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης τώρα τον παρεμποδίζουν ή μάλλον του επιβάλλουν μια λογοκρισία στην ενημέρωση της κοινή γνώμης της Αλβανίας για τα προεδρικά του καθήκοντα, πράγμα που είναι όχι μοναδικό για μένα, αλλά όταν ένας πρόεδρος, ένας αρχηγός κράτους το αναφέρει αυτό, είναι νομίζω ανησυχητικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να εργαστούν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Αλβανία. Και τέλος, ε, σχετικά για τις διοργανικές σχέσεις, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οι ισχυρισμοί του Πρωθυπουργού σχετικά με το δίθεν πραξικόπημα όπου ο Γενικός Εισαγγελέας, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και ο πρόεδρος ο ίδιος ενεπλάκησαν ήταν ε, κάτι που θίγει την αξιοπιστία της χώρας και θα πρέπει να εργαστούμε ούτω ώστε στο μέλλον να προλάβουμε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση. Και η τελική μου παρατήρηση, ναι, είναι ε, ουσιαστικό να, να μιλούμε με μία φωνή ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και εδώ θα ήθελα να πω ότι ήμασταν αρκετά κοντά εμείς όλη αντιπροσωπεία ε, για στην δήλωση της Σοσιαλιστικής Ομάδας για συνεργασία με τον πρόεδρο Μπερίσα για να, για να υπάρξουν οι κανόνες ε, και η εφαρμογή των 12 προτεραιοτήτων κλειδιά και στη μέση αυτής της διαδικασίας λάβαμε την δήλωση του κυρίου Ντόλ ο οποίος σε μια φράση είπε ότι Έντι Ράμα είναι ψυχικά άρρωστος. Δεν θέλω να σχολιάσω τα όσα είπε ο κύριος Ντόλ, αλλά οποιαδήποτε παρόμοια δήλωση όταν γίνεται είτε από το σοσιαλιστή ή από το ΕΛΚ είναι κάτι το καταστροφικό και θα πρέπει να παρεμποδίσουμε στο μέλλον ε, τέτοιες στάσεις, τέτοιες δηλώσεις αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την διαδικασία που βρίσκεται τώρα στα πρώιμα στάδια ε, που είναι κάτι το ευάλωτο ε, που δεν ξέρουμε αν θα διαρκέσει. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα πρέπει να μιλάμε με μία φωνή για να υποχρεώσουμε τις δύο πλευρές να συνεργαστούν προς όφελος της Αλβανίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Και η τελική μου παρατήρηση είχαμε μια εξαίρετη συνάντηση με τη νέα ελίτ στην Αλβανία, τους φοιτητές της πολιτικής σχολής που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους με την ε, συμπεριφορά των πολιτικών ηγετών. Εξέφρασαν την ελπίδα τους και είπαν ότι η Αλβανία αξίζει ένα καλύτερο μέλλον, να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τους ηγέτες της Αλβανίας, αλλά και για την κοινωνία της Αλβανίας στο σύνολό της. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Κασίν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ήμουν παρόν στα τύρανα στην συνάντηση, αλλά παρόλα αυτά μου ζήτησαν οι συνάδελφοι πρώτα ο Στάλι ο οποίος ήταν εκεί εκ μέρους της πολιτικής μου οικογένειας και το προσωπικό της γραμματείας να αρχίσω ευχαριστώντας τον πρόεδρό μας, τον Έντουαρτ Κούκαν, ο οποίος όντως εργάστηκε σκληρά εκεί, απέδωσε με τέτοιες περιστάσεις, χρειάζεται κανείς να είναι διπλωμάτης. Και ε, θα ήθελα να επενέσω τον τρόπο με τον οποίο να μας ανέφερε την κατάσταση εκεί και λυπούμε αγαπητέ Βίκτορ ε, για τα όσα είπες μόλις τώρα. Δεν υπάρχει ανάγκη να επαναλάβουμε αυτά που είπαν, ε, λέχτηκαν μια φορά και αυτού του είδους οι παρατηρήσεις που διαδίδονται εδώ είναι αντιπαραγωγικές. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στο λαό της Αλβανίας, σε αυτές τις πολιτικές οικογένειες για να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ως, όπως ήσασταν δύο από εσά στις δηλώσεις σας. Πιστεύω ότι αυτά τα μπλοκ έχουν τέτοια σκληρή αντιπαράθεση ώστε οι σημερινοί ηγέτες θα πρέπει να δώσουν περισσότερο χώρο όχι μόνο στον πρόεδρο αλλά και στους άλλους πολιτικούς για να αρχίσουν να αναπτύσσουν περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση για να μπορέσουν ε, να σκεφτούν το μέλλον και όχι να εκδικούνται για το παρελθόν. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τους δύο από εσάς ότι αυτό ήταν ένα βήμα προς τα μπρος, αλλά από ασχετικής απόψεως ήταν πολύ μικρό βήμα και δεν υπάρχει εγγύηση ότι το επόμενο βήμα θα είναι στην ίδια κατεύθυνση και όχι σε διαφορετική. Θέλω να είμαι αισιόδοξο και να πιστέψω ότι τον Ιούνιο κάτι θα συμβεί, αλλά φοβούμαι ότι θα χρειαστούμε περισσότερους Ιούνιους για να έχουμε ε, τις ε, κατάλληλες προϋποθέσεις. Καθήκον μας είναι να δραστηριοποιηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ειλικρινεί και να μην εξαπατούμε τους άλλους, να μην του υποσχεθούμε πολλά, διότι χρειαζόμαστε μια συνέχεια στις θετικές εξελίξεις, αν θέλουμε να επανέλθουμε στο επίπεδο που βρισκόταν ήδη η Αλβανία όταν ε, το, το κράτος ήταν κοντά στο καθεστώς αυτό. Υπάρχει ανάγκη για όλο και περισσότερα μεγάλα βήματα και παρόλο που δεν ήμουν εκεί θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόοδο που επετεύχθη και ακόμα και με αυτή τη μικρή πρόοδο θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να είμαστε θετικοί να ε, δώσουμε κίνητρα στις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ε, και στις άλλες επιλογές. Τα πράγματα δεν είναι μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ ε, λύσεις που θα πρέπει να προωθήσουμε στην Αλβανία αν θέλουμε να έχουμε περισσότερη πρόοδο. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Ψωμόπουλο. Τρεμόπουλο. Ήμουν μέλος της ε, Επιτροπής που επισκεφθήκαμε την Αλβανία και είδαμε όλους ε, αυτούς που ανέφερε και ο κύριος Κούκαν, ο οποίος ε, χειρίστηκε πραγματικά με διπλωματία τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εκεί. Θα εστιάσω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει μια αρνητική παράδοση, μια παράδοση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, που πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι φυσικά χωρίς τη συνεργασία των ε, κομμάτων. Υπάρχουν ε, βασικοί τομείς που εγείρουν ανησυχίες όπως η περίθαλψη και η χρηματοδότηση των κομμάτων που πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και να εξυπηρετεί την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα που έχουν οργανωθεί και μπορούν να επηρεάζουν τις εξελίξεις και την πολιτική ζωή. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στρατηγικής για να αντιμετωπιστεί και η έλλειψη διαφάνειας και η διαφθορά και οι τακτικές της. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς δεν εκδικάζονται. Χρειάζεται λοιπόν μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της δικαστικής εξουσίας της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το μεταναστευτικό, το τράφικινγκ, τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων, τον ε, έλεγχο και την πολιτική πίεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος πραγματική στην προστασία του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων και στα θέματα περιουσίας. Και ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για να αντιμετωπιστεί η άνοδος των εθνικιστικών και αλυτρωτικών απόψεων και κινημάτων, ιδιαίτερα στη νεολαία. Τι έχουμε όμως σήμερα εκεί, σε αυτή τη χώρα που είναι διχασμένη και σε μια βαθιά αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Έχουμε την επιστροφή μετά από αρκετό καιρό της αντιπολίτευσης των σοσιαλιστών και τη διάθεση να συμμετέχουν για να καλυφθεί το κενό που χάθηκε όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Τη στιγμή λοιπόν που επανέρχεται στη Βουλή και φαίνεται να ηρεμεί κατά κάποιο τρόπο η πολιτική ζωή εν ώψη του κοινού στόχου έχουμε παρεμβάσεις πολιτικών στελεχών. Ακριβώς σε μια στιγμή σαν να θέλουν κάποιοι να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Αυτές οι παρεμβάσεις που ήδη ακούστηκαν εδώ μέσα δημιούργησαν εντελώς αρνητικό κλίμα στην επαφή μας με τον ηγέτη των σοσιαλιστών. Δεν βοηθούν λοιπόν αυτές οι παρεμβάσεις με ανεπίτρεπτους μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς και μάλιστα από σοβαρά στελέχη εδώ του Ευρωκοινοβουλίου εναντίον του ηγέτη των σοσιαλιστών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και με αυτή την πλευρά αυτό που ο κύριος Κούκαν ανέφερε ως ανάγκη για κοινή γλώσσα και όχι λανθασμένα μηνύματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εξηγήσαμε στον πρόεδρο των σοσιαλιστών ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ένα πράγμα. Ακόμη και στα ίδια τα κόμματα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό έγινε κατανοητό και προσπαθήσαμε να κλείσουμε αυτά τα τραύματα που στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου έχουν δημιουργήσει. Ελπίζουμε αυτά να μην ε, έκλεισαν προσωρινά τα ζητήματα και πραγματικά στα βασικά σημεία, πέρα από τις διαφορές τους, τα δύο μεγάλα κόμματα και οι ηγέτες να μπορέσουν να επιτύχουν αυτή την πρόοδο που θέλουμε για να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας που να παίξει έναν πραγματικά σταθεροποιητικό ρόλο και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι όσοι ήθελαν να πάρουν τον λόγο τον πήραν. Τελειώνουμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο, 13. Έκθεση σχετικά με την αντιπροσωπή εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε στην Ικαράγουα ευευκαιρία των γενικών εκλογών της 6ης Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία πήγε στην Ικαράουα 3 με 8 Νοεμβρίου. Θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο της αντιπροσωπείας αυτής, την κυρία Γιάλα Σάντερ, για να μας ε, παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Θέλω να παρουσιάσω στην Επιτροπή αυτή την έκθεση της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε την τιμή και την ευκαιρία, που είχα μάλλον την τιμή και την ευκαιρία να προεδρεύσω εγώ. Ήταν ε, όντω το ταξίδι αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και καρποφόρο. Όντω οι εκλογέ έγιναν στι 6 Νοεμβρίου για πρόεδρο και αντιπρόεδρο τις χώρες από την μια μεριά και από την άλλη μεριά τους βουλευτές εθνικούς και περιφερειακούς όπως επίσης και στο Παρλαφέν. Υπήρξαν όμως κάποιες επιπλοκές από πριν πρώτα απ' όλα. Ήδη από το 2008 όπου είχαμε τοπικές και περιφερειακές εκλογές και εκεί εντοπίστηκαν ε, μέχρι και απάτες. Γι' αυτό και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά την άμεση βοήθεια στην Ικαράγουα που ήταν να σταματήσει τη βοήθεια αυτή. Λίγο πριν τις εκλογές βλέπετε ο πρόεδρος Ορτέγα υπέβαλε και πάλι την υποψηφιότητά του για την Προεδρία παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Σύνταγμα της Νικαράγουα απαγορεύει δύο διαδοχικές θητείες. Το Ανώτατο Δικαστήριο ε, δέχτηκε την υποψηφιότητα αυτή που καταρχήν είναι αντισυνταγματική και έτσι τελικά οι εκλογές αυτές ξεκίνησαν με αυτή την παραφωνία. Τα υπόλοιπα κόμματα τώρα υπό τη μορφή συμμαχιών αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις εκλογές γιατί η κατάσταση όσον αφορά τα κόμματα στην Ικαράγουα είναι τέτοια που λέει ότι αν δεν συμμετέχουν στις εκλογές τότε χάνουν το δικαίωμα να αποτελούν κόμμα. Πέρα λοιπόν από το θέμα της υποψηφιότητας στην Προεδρία του Ντανιέλ Ορτέγα υπήρξε και ένα άλλο πρόβλημα με το ανώτατο εκλογικό όργανο της Νικαράγουα, της Νικαράγουα που είναι το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο. Αυτό έπρεπε να ανανεωθεί. Μετά τα προβλήματα και την απάτη για τις εκλογές του 2008 έπρεπε να αποχωρήσουν κάποιοι δικαστές και να ανανεωθούν. Ε, έκανε ο πρόεδρος χωρίς να περάσει από την Εθνική Συνέλευση ανανέωσε τη θητεία τους εκείνος με ένα διάταγμα. Οπότε τελικά ένα νότατο εκλογικό συμβούλιο που είναι το νότατο όργανο που οργανώνει τις εκλογές και που έχει μεγάλη επιρροή στα κόμματα, μια που δεν υπάρχει άλλος ε, εκλογικός νόμος, τελικά αποτελείται από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ε, οργανώσει και τις προηγούμενες εκλογές τις οποίες είχαν εντοπιστεί οι απάτες, το 2008 δηλαδή. Η αντιπροσωπεία μας κάποια στιγμή το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει πολιτική πρόσκληση για να πάνε παρατηρητές, στις 17 Αυγούστου, όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός για, όπως το ονομάσαμε, συνοδεία στις εκλογές, ο πρόεδρος Ορτέγα έκανε μία δήλωση με την οποία τελικά ε, μας υποδεχόταν ευχαρίστως έλεγε ως παρατηρητές και ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και πλήρη ελευθερία κινήσεων. Υπήρξε ένα μνημόνιο κατανόησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Νότατο Συμβούλιο και με την κυβέρνηση και έτσι τελικά οι κανόνες βάσει των οποίων θα διεξάγονταν ε, η παρατήρηση αυτή των εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν κάτι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες. Τον Οκτώβριο αποφασίστηκε η αντιπροσωπεία αυτή, η αποστολή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των όσων ανέφερε το, μνημό, Μνημόνιο Κατανόησης ήταν ο κύριος Ρουίς Γιάννεθ και άλλοι 90 παρατηρητές οι οποίοι κάλυπταν ε, όλη τη χώρα έτσι ώστε παντού στη χώρα να υπάρχουν ομάδες. Είχαν προετοιμαστεί από νωρίτερα πολύ καλά και έτσι μπορούσαν να παρατηρήσουν τις εκλογές πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν τον Νοέμβριο η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία προσθέθηκε στους υπόλοιπους παρατηρητές Πήγε με έξι συναδέρφους και την γραμματεία, η οποία βοήθησε πολύ και θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία της, προκειμένου να φέρουμε σε πέρα στη δουλειά μας κάτω από τις καλύτερες δυνατόν ε, συνθήκες. Οι συνάδελφοι είναι εδώ, είναι η κυρία Αναγόμες, που είναι, δεν βλέπω άλλους, ο κύριος Κασμάρη, ο κύριος Σόνικ, ο κύριος Λόπεθ Άγγιλαρ, ο κύριος ε, Χισνούσικ και η κυρία Γκρέσε. Όλοι εμείς μαζί λοιπόν, λίγες μέρες πριν τις 6 Νοεμβρίου, είχαμε επαφές και με τον πρέσβη, τον κύριο Μέντελ Γκόλστεν, ο οποίος μας βοήθησε και μας έδωσε ό,τι πληροφορίες θέλαμε, ό,τι μέσα χρειαζόμασταν, τα, μας τα διέθεσε, αλλά και με τους πρέσβεις από διάφορες χώρες μέλη, σε δύο γύρους, όταν πήγαμε και πριν φύγουμε. Δύο φορές δηλαδή συναντηθήκαμε μαζί τους για να ακούσουμε τη γνώμη τους για τα όσα έγιναν. Πριν από τις εκλογές λοιπόν ε, συναντηθήκαμε και με τους διάφορους υποψηφίους και με τον Τανιέλ ε, Ορτέγα θελήσαμε να συναντηθούμε αλλά δεν μπορέσαμε και με τον Νότατο Εκλογικό Συμβούλιο το οποίο επίσης μας ενημέρωσε και σχολιάσαμε με τον Πρόεδρο και τους δικαστές τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί όσον αφορά ε, τις ε, επιτροπές εκλογικές στα διάφορα εκλογικά κέντρα και άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα με τους δικαστές, όπως είπαμε, στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Ε, και εκείνοι είχαν αναγνωρίσει ότι τα ψηφοδέλτια ήταν τα πολύ περισσότερα από αυτός που μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι και οι νεκροί είχαν ψηφίσει. Και ότι ε, όσοι δεν ήταν στους εκλογικούς καταλόγους παρόλα αυτά μπορούσαν να προσθέσουν το όνομά τους και να ψηφίσουν. Δηλαδή υπήρχε μια τεράστια ευελιξία για να το πούμε έτσι. Το αναγνώρισε αυτό δηλαδή και το ίδιο το Νότατο Εκλογικό Συμβούλιο. Συναντηθήκαμε και με τους εθνικούς παρατηρητές επίσης, αυτοί οι οποίοι δεν πήραν την άδεια γιατί το Νότατο Εκλογικό Συμβούλιο δεν ε, διαπίστευσε όλους όσοι το επιθυμούσαν, ε, του θεωρούσε ότι δεν ήταν ευνοϊκά διατεθειμένοι, δεν ήταν συμπαθητικοί και δεν τους το επέτρεψε. Εμάς όμως μας διευκόλυναν, αυτό πρέπει να το πω. Μας βοήθησαν πολύ. Την ημέρα των εκλογών τώρα ήμασταν τέσσερις ομάδες στην Μανάγουα, στο... Λέω, στη Γρανάδα και πρέπει να το αναγνωρίσω, είναι κάτι θετικό για τις εκλογές αυτές, ότι δεν υπήρξε βία η κατάσταση βίας που είχαμε διαπιστώσει σε άλλες εκλογές δεν υπήρξε αυτή τη φορά. Είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίσαμε και εμείς και το αναγνώρισαν και όλοι. Πέρα από τα προβλήματα ε, διαπίστευσης ε, κλπ. Δεν υπήρξαν προβλήματα βίας. Οπότε την ημέρα των εκλογών μπορούμε να πούμε ότι ο πληθυσμός πήγε να ψηφίσει εν ελευθερία. Βέβαια είναι κάτι διαφορετικό το κατά πόσες συνθήκε ήταν οι καλύτερες δυνατόν για να ε, ψηφίσουν. Σας είπα τα προβλήματα με τους δικαστές, με τους εκλογικούς καταλόγους και με την ε, παρατήρηση από τους εθνικούς παρατηρητές που δεν ε, μπορούσε να γίνει γιατί δεν πήρα διαπίστευση για την παρατήρηση των εκλογών. Ήμασταν εκεί μέχρι που έκλεισαν τα εκλογικά κέντρα και κάναμε την πρώτη μας έκθεση, δηλαδή τόσο η αντιπροσωπεία μας Συναντηθήκαμε πολλές φορές και με τον κύριο Γιάννη, τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι προσπαθήσαμε να συμπληρώσουμε και εμείς την ίδια γραμμή πάντα με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και εμείς ήμασταν κριτικοί. Είπαμε ότι ναι, μεν με ελευθερία ψήφισαν οι πολίτες, αλλά μιλήσαμε και για τα προβλήματα που υπήρχαν. Μέσα στις 24 ώρες είχαμε τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα, αλλά ήδη είχαμε εντοπίσει παρατυπίες. Αυτό το οποίο τόσο η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η δικιά μας αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίσαμε ότι το μέτωπο των Σαντινίστας κέρδισε τις εκλογές αυξάνοντας βέβαια κάπως περισσότερο το ποσοστό από πριν, αλλά και αντιπολίτευση, η UN Fleet, ε, με τον ε, πρόεδρο, τον Κουαντέα, και αυτοί προχώρησαν. Και ο Αρνόλντο Αλεμάν και ο Φάβιο Καδέα τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε απάτη, τουλάχιστον η δικιά μας αντιπροσωπεία δεν λέει ότι υπήρξε απάτη, δηλαδή τον, τα ονόματα άλλαξαν οι σταυροί, όχι. Ο πρόεδρος πάντως ο Ντανιέλ Ορτέγα του FSLN πράγματι κέρδισε τις εκλογές. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως ήταν ότι η διεξαγωγή των εκλογών δεν έγινε χωρίς παρατυπίες και ότι η διαφάνεια, η παρατήρηση, ο έλεγχος, η παρακολούθηση των εκλογών έγινε μέσα σε περίπλοκες και δύσκολες συνθήκες. Και μάλιστα αφού γυρίσαμε διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν κάποιες ε, αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Με πέντε νεκρούς μάλιστα. Σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Εκεί όπου ε, ιστορικά ε, υπήρχαν διαφορές με την κυβέρνηση. Οι ευρωβουλευτές ε, συντάξαμε λοιπόν μια έκθεση. Λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, να έχει τα οριστικά αποτελέσματα. Και επίσης ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε εκτός από τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς θα ξεκινήσει να δουλεύει η συνέλευση. Να δούμε δηλαδή με τις δαγματικές αλλαγές που ο πρόεδρος Ορτέγα ε, θα κάνει, έχει μεν ε, αρκετή πλειοψηφία, αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να το κάνει από μόνος του, θέλει να το κάνει μέσα από την συνέλευση. Αυτό πρέπει να δούμε, αν θα το κάνει όντω έτσι. Και αν το δημοκρατικό παιχνίδι θα παιχτεί σωστά, παρά την ε, σημαντική πλειοψηφία που έχει ο πρόεδρος Ορτέγα. Ιδίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών τώρα μετά τη Λισαβόνα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τις αρμοδιότητες μας αυτές για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να πάρουμε αποφάσεις ανάλογα με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, έτσι ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η δημοκρατία στην Ικαράγουα. Λοιπόν, είναι μια χώρα φτωχή, από τις πιο φτωχές αυτού του τμήματος του ημισφαιρίου. Πλήττεται από φτώχεια. Παρ' όλα αυτά είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα και τα σχέδια του FSLN έδωσαν μια δυναμική ανάπτυξη του 4% στη χώρα. Βέβαια η ανάπτυξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να ψηφίσουν πολύ το FSLN, εννοείται. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες που και εμείς επικρίνουμε και αναγνωρίζονται και έχει να κάνει με τα χρήματα που δίνει η Βενεζουέλα 500 εκατομμύρια το χρόνο που δεν περνάνε από ό,τι φαίνεται από τον προπολογισμό και από τον ε, δημοκρατικό έλεγχο προπολογισμού. Οπότε πρέπει να δούμε ποια είναι η δυνατότητα που έχει το FSLN να προχωρήσει με προγράμματα ανάπτυξης στο μέλλον για τους κατοίκους Θέλουμε δηλαδή από τη μια να δούμε ανάπτυξη και δυναμική θετική στην Ικαράγουα από την άλλη μεριά όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάλογος και πραγματική δημοκρατία στην συνέλευση, να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Μήπως είναι αυτή μια μεγάλη αδυναμία. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Και η δημοκρατική σταθερότητα στην συνέλευση να διατηρηθεί και ο πρόεδρος Ορτέγα να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία αυτή θετικά και όχι για αντισυνταγματικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Γιάλα Σέντες. Η κυρία Δίνω Γκόμες. τώρα τον λόγο στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, Νομίζω ότι η αντιπροσωπεία ε, διευθύνονταν πολύ καλά από την ε, συναδελφό μας, την κυρία Γιάλα Σέρα και θα ήθελα να αποδώσω φόρο ε, στην εργασία της και να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που ήταν στην, στο ταξίδι αυτό και την γραμματεία του Κοινοβουλίου. Άμεθα πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, όπως η Νέσ εξήγησε δεν υπήρξε άμεση νοθεία, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και δίκαιες αυτές οι εκλογές. Δεν χρησιμοποίησαμε όμως αυτή την ορολογία. Θα έπρεπε να πούμε εδώ ότι δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Και όπως λέχθηκε υπήρξαν πάρα πολλές παρατυπίες. Ε, βεβαίως ε, λήφθηκε η απόφαση βάσει του συντάγματος να αναθεωρηθούν όλες οι διαδικασίες ε, ούτως ώστε ο κύριος Ορτέγκα να μπορέσει να ξαναπαρουσιαστεί άλλη μία φορά. Μια κατάσταση κάπως γελία και οι εκπρόσωποι ε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν ήταν ε, ε, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αλλά είχαν οριστεί από το κόμμα της εξουσίας. Βλέπετε λοιπόν πώς υπήρξε χειραγώγηση των εκλογών. Τις ημέρες πριν από τις εκλογές ένα από τα κανάλια τηλεόρασης είχε έναν παρουσίασε έναν επίσκοπο που ε, υποστήριζε τον Ορτέγκα, που παρότρινε τον κόσμο να ψηφίσει υπέρ του Ορτέγκα. Και νομίζω ότι είναι όνειδος να βλέπει κανείς μια χώρα με εξαιρετικό πληθυσμό, με την ιστορία που έχει, είναι ντροπή να βλέπει κανείς την παρούσα κατάσταση που βρίσκεται στα χέρια μιας ολιγαρχίας που κρατιέται στην εξουσία Πρέπει να πω ότι είναι εντυπωσιακό να δει την δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, εξεπλάγει από την δραστηριότητα των οργανώσεων, των οργανώσεων για παρατήρηση των εκλογών, οργανώσεις οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές που ασχολήθηκαν με εκλογές εκτός Νικαράγουας. Επίσης, Ε, θα πρέπει εμείς να μην εγκαταλείψουμε την Ικαράγουα, αλλά να αποδώσουμε περισσότερη σημασία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στην Ικαράγουα. Ο πρόεδρος Σορτέγα ε, ακολουθεί το δικό του σχέδιο για να παραμείνει στην εξοχή. Ευχαριστώ, Γκάλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, της Αποστολής ε, για την έκθεσή τους και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ διδακτικό για όλους. Τα όσα είπε η Αναγκόσμες ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη χώρα αυτή, με τους πολίτες της και να μην ασχολούμε με την ευζοία και ευημερία του Προέδρου. Τον γνωρίζουμε από την εποχή που υπήρχαν τα δύο μπλοκ Ανατολής και Δύσης τη δεκαετία του 80 όταν για πρώτη φορά κέρδισε την νίκη με το κίνημά του και είπε τότε η Επανάσταση κέρδισε και είμαστε στην εξουσία αντετέρναμ. Όταν αντελήφθη ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι έτσι, παρουσιάστηκε με δημοκρατικό πρόσωπο, αλλά έχω πράγματι την εντύπωση ότι και ε, ε, γίνεται το ίδιο όπως και στην Αφρική όταν ε, το Σύνταγμα δεν, επιτρέπεται, δεν επιτρέπει νέα υποψηφιότητα, χειραγωγεί κανείς το Σύνταγμα για να παραμείνει στην εξουσία κάθε φορά που διαπιστώνουμε τέτοια φαινόμενα πρώτων εκλογών θα έπρεπε απλώς να πούμε ότι στις χώρες αυτές δεν θα πρέπει πλέον να πηγαίνουμε στις χώρες ως παρατηρητές διότι υπάρχει κατάφορος χειραγώγηση ανεξάρτητα του, του, του του τι συμβαίνει στη συνέχεια. Ακόμη και αν μετά διαπιστώνουμε νοθείες, απάτες, εδώ δεν ήταν η περίπτωση, αλλά αν στην αρχή ε, τα στοιχεία είναι νοθευμένα, αν παρουσιάζεται ως υποψήφιος κάποιος που δεν έχει το δικαίωμα, θα έπρεπε εμείς να είμαστε συνεπείς και να πούμε ότι ο ελάχιστος κανόνας δεν τηρείται και θα πρέπει να το λέμε δυνατά. Ίσως θα έπρεπε απλώς να πούμε ότι ορισμένα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ευχαριστώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και την Αγιάλα ε, Σέντερ για την έκθεση που ήταν πλήρης. Και τώρα περνάμε στο σημείο 14 η έκθεση σχετικά με την αντιπροσωπεία εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γενικέ εκλογές 28 Νοεμβρίου και που βρισκόταν επιτόπου από τις 26 στι 30 Νοεμβρίου. Θα δώσω τον λόγο στην Μαριάν Νεντελ που ήταν επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Παρατηρητών για τις εκλογές του 28 Νοεμβρίου και του κ. Περέλο που ήταν επικεφαλής ε, της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε αυτή την ίδια χώρα. Πρώτα απ' όλα η κυρία Νέτσαβά και μετά ο κύριος Περέλο Ροντρίγκερς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περέλο ε, για την ε, διεύθυνση της αποστολής ε, που πήγε στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με την ευκαιρία των εκλογών, των βουλευτικών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιελάμβανε 140 παρατηρητές που αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα στις 11 επαρχίες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι αυτό που αποτελεί μέρος της μεθοδολογίας μας είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία, αλλά είναι μια ε, μεθοδολογία μακροπρόθεσμη. Οι παρατηρητές μας που από τις 18 Οκτωβρίου αναπτύχθηκαν στην επικράτεια, παρακολούθησαν την προεκλογική στρατεία, τα διάφορα στάδια ε, μέχρι την ημέρα των εκλογών και μετά με την, ε, τα αποτελέσματα η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έκθεση της οποίας θα παρουσιάσω στην Επιτροπή, βασίζονται σε άμεσες παρατηρήσεις από τους παρατηρητές μας. Θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να πούμε ότι η έκταση της αποστολής μας είναι αρκετά περιορισμένη. Οι διαπιστώσεις μας περιορίζονται στις αστικές περιοχές. Δεν έχουμε Άμεσε παρατηρήσει από τι αγροτικές περιοχές, εξού η σημασία της συνεργασίας που είχαμε από την αρχή με τις διεθνεί και εθνικές αποστολέ, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο ε, σημαντικό και θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη συνεργασία διότι όταν μας κατηγορούν ότι ο αριθμός των παρατηρητών στις χώρες ε, δεν αρκούν για όλα τα εκλογικά τμήματα και στην ε, περίπτωση του Κονγκό το μέγεθος της χώρας και ότι έχει, είχε 63.000 εκλογικά τμήματα και δεν μπορούσαμε να καλύψουμε, μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό με την συνεργασία με διεθνείς και εθνικές αποστολές επιστολές παρατηρητών. Θα ήθελα να σας πω ποιο ήταν το πλαίσιο των εκλογών 2011 σε σχέση με το 2006. Είναι οι δεύτερες εκλογές ε, για την ε, εδραίωση της δημοκρατίας ε, στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Αυτή τη φορά η ηγεσία ήταν κογκολέζικη. Μπόρεσε να συμβάλλει οικονομικά ε, σε 80-90% αυτή τη φορά ήταν η ΦΥΝΗ, η Εθνική Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή που ήταν επιφορτισμένη με την οργάνωση και την διαχείριση αυτών των εκλογών. Αυτές οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από σημαντικά συνταγματικά, συνταγματικές διαφορές και ε, αυτό που αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση μας ε, και είναι η κινητοποίηση ορισμένων περιφερειών, ορισμένων οχυρών που αρκούσαν ε, για την εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχαμε τέσσερα στάδια. Όσον αφορά την οργάνωση αυτών των εκλογών, υπενθυμίζω ότι ήταν σημαντικές προκλήσεις ε, οικονομικές, ε, επιμελητίας και υλικές βλέπουμε ότι δεν, ε, ο κατάλογος δεν ήταν αντικείμενο ε, συμβίβασμου. Ε, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπόρεσε με τη σειρά της να επιτύχει την έκθεση που, που είχε κάνει το ξεκαθάρισμα το εκλογικό. Και αν επισύρω την προσοχή πάνω στο θέμα αυτό είναι επειδή έχουν, υπήρξαν πολλές φήμες, εικασίες για τον ε, αριθμό των επικαλύψεων ε, σε αυτό το μητρό. Ε, περάσαμε σε 119.000 από το φινί που είναι αντικείμενο κριτικών. Δεύτερον, όσο αφορά την χαρτογράφηση των εκλογικών τμήματων, είναι σαφές για μας που ότι θα πρέπει σαφώς να υπάρχει μια σαφής τέτοια χαρτογράφηση, ούτως ώστε τα πολιτικά κόμματα να μπορέσουν να οργανωθούν, να δουν πού θα στείλουν παρατηρητές την ημέρα των εκλογών. Σχετικά με την ανάπτυξη υλικού στα διάφορα εκλογικά τμήματα, παρατηρήσαμε με την πάροδο των εβδομάδων ότι η Θηνή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, αλλά αυτό που παρατηρούμε εξ αρχής είναι μια έλλειψη επικοινωνίας και διαφάνειας στην εργασία αυτή την προεκλογική πράγμα που τροφοδοτεί κριτικές οι οποίες δεν αρκούνται μόνο στη σύνθεση της Φίνη αλλά στον τρόπο επικοινωνίας της και στις προσπάθειες που κατέβαλε για την οργάνωση των εκλογών. Δεύτερον, σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία, η οποία για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ισορροπία στο μέτρο που η πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν ίση για όλους οι υποψήφιους. Μετά την ανάλυση που κάναμε βλέπουμε ότι 80% της πρόσβασης ήταν, επιφυλασσόταν για τον απερχόμενο πρόοδο και για την, και είχαμε ε, την ανώτερη δικαστήριο για τα οπτικοακουστικά που παραμένει ένα κενό κέλυφος. Δεύτερο πράγμα, επισύρουμε την προσοχή πάνω στην χρησιμοποίηση των πόρων του κράτους και την έλλειψη ενός νόμου για την χρηματοδότηση των κομμάτων. Ε, αυτά τα δύο κενά δημιούργησαν ανισότητες αρκετά σημαντικές στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Παρατηρώ επίσης τον ρόλο των πάρα πολύ αμφιλεγόμενων των δίκητων που οι περισσότεροι ήταν υποψήφοι και καμιά φορά η διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο λειτουργήμα και στο πολιτικό του υποψηφίου σε εκλογές, αυτή η διάκριση δεν ήταν και ο διαχωρισμός δεν ήταν σαφής. Είχαμε τον ρόλο των θετικών όμως διαφόρων πλατφορμών που επέτρεπαν στις πολιτικές δυνάμεις να έχουν διάλογο και να αμβλύνουν ε, τις εντάσεις. Υπήρχε το φόρουμ των πολιτικών κομμάτων ε, που συνεδρίασε τρεις φορές, αλλά στο επίπεδο των περιφερειών είδαμε ότι εκεί όπου υπήρχε ένα τέτοιο βήμα δηλαδή τα, οι επιτροπές μεσολάβησης υπό την αιγίδα της Αμμονισκό μπόρεσαν να ε, αμβλύνουν την ένταση. Σχετικά με την ημέρα των εκλογών, αυτό που παρατηρήσαμε είναι μια ισχυρή κινητοποίηση και επαγρύπνηση των ε, πολιτών που είχαν ένα έντονο πολιτικό αίσθημα. Την ημέρα των εκλογών ε, πρέπει, έπρεπε κανείς να είναι προσεκτικός και να μιλήσει για αντιθέσεις στην κατάσταση. Υπήρξαν εκλογικά τμήματα που άνοιξαν στην ώρα τους, που ήταν καλά εξοπλισμένα και λειτουργικά, αλλά αυτό δεν μας κάνει να ξεχνούμε τα εκλογικά τμήματα όπου η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ακόμη και χαοτική λόγω έλλειψης ελεγχόμενης οργάνωσης, πράγμα που οδήγησε σε αρκετές εντάσεις σε ψηφοφόρους που δεν βρίσκαν τα ονόματά τους στους καταλόγους και εκεί με την προσοχή πάνω στο γεγονός ότι το 2006 η Ευρωπαϊκή Αποστολή έκανε συστάσεις σχετικά με τον κατάλογο αυτών που είχαν παρελειφθεί. Αυτή την φορά βλέπουμε ότι αν το 2006 ήταν 8% αυτοί που είχαν παραλυφθεί, αυτή τη φορά 17% είχαν παραλυφθεί και μπόρεσαν να εγγραφούν χάρη σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό μας παραπέμπει στο θέμα του εκλογικού μητρώου. Όσον αφορά την ημέρα των εκλογών, το γεγονός ότι ε, τα δελτία δεν υπήρξαν αρκετά γέρος, δημιούργησε εντάσεις. Επίσης, η θέση των γυναικών που θα πρέπει να ενισχυθεί σε σχέση με το 2006 δεν υπήρξε πρόοδος στον τομέα αυτό, δεν υπήρξε καμία υποψήφια γυναίκα για τις προεδρικές εκλογές και ο αριθμός των γυναικών υποψηφίων στις βουλευτικές ήταν το ίδιο ποσοστό με το 2006, γι' αυτό γίνεται έκκληση για να υπάρξει η τήρηση της αρχής της ισότητας που υπάρχει στο Σύνταγμα σχετικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το τελευταίο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, οι παρατηρητές μας μπόρεσαν να επισκεφθούν τα τοπικά κέντρα ε, ε, για τα αποτελέσματα των εκλογών και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ε, παρατυπίες και κενά και διαπιστώσαμε την έλλειψη στοιχείων κλειδιών που εγγυώνται ε, την νόμιμότητα και που μπορούν να θίξουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που για μας ήταν στη θέα προστασίας. Αφενός η παρουσία διαφόρων εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, ε, ε, πάρα πολλές φορές όμως δεν έγινε η δεχτή η παρουσία τους. Κιντσασά, Κατάγκα, η επαρχία η Ανατολική. Δεύτερο στοιχείο στη θεοπροστασίας για μας είναι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Το άρθρο 70 του εκλογικού νόμου. Αυτό δεν τηρήθηκε αμέσως παρατηρούμε περιπτώσεις όπως σε αντίφαση με τον εκλογικό νόμο το γραφείο της ΣΕΝΗ ζήτησε να μην αναρτηθούν αμέσως τα αποτελέσματα και να σταλούν πρώτα στο έδρα της ΣΕΝΗ για να ελεγχθεί η συνεκτικότητα ε, και στην Γκόμα, Μάντακα, Μαζαγκουρού, Κιντσασάκη, Σαγκανή και Λουμουμπασί διαπιστώθηκαν τέτοιες ελλείψεις. Τρίτο στοιχείο για το Εθνικό Κέντρο Επεξεργασίας των Αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το όργανο το οποίο ε, βάζει μαζί τα αποτελέσματα. Εδώ ούτε από τα πολιτικά κόμματα, ούτε κανένα παρατηρητή δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο για μα είναι κεντρική σημασία είναι ε, από το κάθε εκλογικό κέντρο το αποτέλεσμα τα αποτελέσματα δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται προς το παρόν είναι ότι τα πρακτικά αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν είναι ε, μηχανογραφημένα και περιμένουμε πάντα ε, τα πρακτικά από το κάθε εκλογικό κέντρο και είναι και ορισμένα τα οποία δεν έχουν ληφθεί καν υπόψη στις εκλογές αυτές. Εμείς υπολογίσαμε 4.875 πρακτικά, τα οποία δεν μετρήθηκαν και είναι 1,6 εκατομμύρια εκλογής δηλαδή, ε, τον οποίων η ψήφος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Και θέλω να τελειώσω με ένα τελευταίο σημείο το οποίο μας κάνει να αναρωτιόμαστε και η επιστολή, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει ήδη δηλώσει, είναι το ανώτατο δικαστήριο. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκφράσει τις ανησυχίες της λέγοντας ότι κατά την εκλογική, προεκλογική εκστρατεία δεν μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση στους υποψήφιους και τις αποφάσεις σχετικά με τους υποψήφιους αυτούς. Δεν τις έχουμε δει ακόμα. Το ανώτατο δικαστήριο είναι το όργανο το οποίο κανονικά διαχειρίζεται όσο γίνεται καλύτερα ε, όλους τους υποψηφίους και θα θέλαμε να είχαμε μια ακρόαση μετά την ακύρωση των αποτελεσμάτων για τον κύριο Καμερέ. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να δούμε το περιεχόμενο, πώς ελήφθη η απόφαση αυτή. Διαπιστώνουμε όμως δυστυχώς ότι το ανώτατο δικαστήριο δεν χαίρει της εμπιστοσύνης του λαού, ενώ θα έπρεπε κανονικά. Οπότε η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα υπογραμμίζει τα στοιχεία αυτά και σας υπενθυμίζω ότι οι προεδρικές εκλογές είναι ένα τμήμα μόνο, γιατί υπάρχουν και γενικές εκλογές. Οπότε αν επιτρέπουμε στους αυτούς μας να υπογραμμίζουμε τα στοιχεία αυτά, είναι γιατί αυτά τα στοιχεία ε, δείχνουν ελλείψεις και αν δεν υπήρχαν θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια και για τις γενικές εκλογές έτσι ώστε οι πολίτες της χώρας να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι τα αποτελέσματα που τους ανακοινώνουν είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ταξίρα, πραγματικά ήταν πολύ πλήρη η παρουσίασή σα. Ο κύριο Σοπερέ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όσοι έχουν αντισταθεί και βρίσκονται ακόμα εδώ, δεν θα τους ε, δυσκολέψω εγώ περισσότερο τη ζωή μακρηγορώντας. Εξάλλου, ο συνάδελφος τα είπε πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως που πρέπει εδώ να σας πω, ότι δεν το λέω από ευγένεια, αλλά πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία, αλλά και την γραμματεία, αλλά και όλους τους παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κυρία Νεντιτσέβα. Η αποστολή αυτή είχε μια δύσκολη δουλειά εξαιτίας της κατάστασης στη χώρα πρώτα απ' όλα και έπρεπε να διακινδυνεύσει μερικά πράγματα για να πάνε τα πράγματα καλά. Αυτό το λέω να το ξέρετε. Τώρα, στο βαθμό που συμμετείχαμε στην αποστολή παρατήρησης των εκλογών και συμφωνούμε με την έκθεση της αποστολής, δεν θα είχαμε πολλά να προσθέσουμε. Μια λεπτομέρεια όμως. Υπάρχουν θετικά πράγματα στη διαδικασία και κάτι αρνητικό. Μερικές φορές είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την διεξαγωγή δεύτερων εκλογών στην ιστορία αυτής της χώρας που είναι περίπου μια ολόκληρη ήπειρος και γίνονται εκλογές αυτές ενώ λείπουν τα πάντα. Υποδομές, αυτό που λέμε εμείς δρόμοι δεν είναι το ίδιο με αυτό που λένε αυτοί οι δρόμοι. Οι ελλείψεις δηλαδή είναι τεράστιες. Μια πόλη με ένα εκατομμύριο κατοίκους όπως είναι η Κινσάσα χωρίς ε, μεταφορές ε, δημόσιες. Είναι φοβερό δηλαδή οι διαφορές που υπάρχουν με αυτά που ξέρουμε εμείς. Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα που αποτελεί ένα ακόμα παράδοξο στον πλανήτη αυτό. Δεν είναι φτωχή χώρα, έτσι, είναι πλούσια χώρα, αλλά με φτωχό λαό. Κάτι το οποίο μας μπερδεύει και εμάς ακόμα. Οι λόγοι βέβαια είναι ιστορικοί και άλλοι πολλοί. Το, ποιο είναι το θετικό, ότι ο κόσμος ήθελε να πάει να ψηφίσει και πήγανε στα εκλογικά κέντρα. Και μιλάω γενικά, γιατί εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις σας τα είπε και η κυρία Νεντετσέβα. Στα εκλογικά κέντρα λοιπόν, βλέπαμε και τον κόσμο που πήγαινε να ψηφίσει ευχαρίστως, αλλά βλέπαμε και ε, τους υπεύθυνου εκεί να θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τα είπε και η κυρία Νεντελτσέβα τα προβλήματα προέκυψαν πότε, μετά, ότι χάθηκαν τόσα ψηφοδέλτια, ότι αυτός που βάζει τα στοιχεία στον υπολογιστή δεν ελέγχεται από κανέναν, μπορεί να αφήσει απ' έξω 10.000. Δηλαδή σε τέτοια πράγματα υπήρξαν ε, προβλήματα. Ήταν εκλογές για τον πρόεδρο. Θα έπρεπε να ήταν απλό. 11 φωτογραφίες, 10 ε, άντρες, μία γυναίκα. Θα έπρεπε να είναι εύκολο. Βλέπει κανείς τη φωτογραφία, από κάτω σημειώνει, τελείωσε. Και το ρίχνει στην κάλπη. Φανταστείτε όμως τι γίνεται όταν έχουμε 20.000 υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές. Στην Κινσάσα 1980 υποψήφοι υπάρχουν για μία θέση. Εκεί το ψηφοδέλτιο θυμίζει η εφημερίδα όπως είναι η Mondo ή η Financial ε, Times με 50 σελίδες. Πού να ψάξει να βρει τη φωτογραφία και αυτούς που θέλει τέλος πάντων να ψηφίσει, να διπλώσει μετά το ψηφοδέλτιο αυτό και να το βάλει στην κάλπη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο είναι να γίνει αυτό το βράδυ με κερί, γιατί δεν υπάρχει πάντα ηλεκτρικό. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, είναι σοβαρό. Γιατί οι υποψήφοι πρέπει να δούμε, δέχονται τα αποτελέσματα. Δεν έγινε όμως αυτό. Οπότε η διεθνής κοινότητα έχει μεγάλο ρόλο να παίξει. Σήμερα υπάρχει ένας καινούριος πρόεδρος στο Κονγκό που έχει υποσχεθεί ε, δυνάμει ασφάλεια κλπ. Αλλά ο άλλος υποψήφιος, ο Κισεκέδη, τι λέει, λέει ότι εκείνο θα αναλάβει μέσα στο στάδιο με τους δικούς του. Οπότε θα έχουμε δύο πρόεδρους. Ένας που επίσημα έχει κηρυχθεί πρόεδρος και άλλος ανεπίσημα. Δηλαδή έχουμε ό,τι συστατικά χρειαζόμαστε για ένα νέο εμφύλιο πόλεμο. Ελπίζω να μην γίνει έτσι και να υπερβάλλω αλλά τα συστατικά υπάρχουν όσο περνάνε οι μέρες, αυτό βλέπουμε. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν πρέπει να τοποθετηθεί. Αναγνωρίζω ότι εδώ σας δίνω την ε, δικιά μου, την ε, προσωπική γνώμη. Προσοχή τι γίνεται με όλες τις ε, επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα αυτή και τι ρόλο παίζουν. Έτσι κι υπάρχει μεγάλη διαφθορά στη χώρα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυτικέ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν λέω ότι έχει άμεση σχέση αυτό με τις εκλογέ, αλλά μπορεί να έχει τη σημασία του. Μην δηλαδή τοποθετηθούμε ανάλογα ο καθένας μας με τα συμφέροντα που μπορεί να έχει στη χώρα αυτή. Σημαντικό είναι να υπάρχει δημοκρατία σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Από εκεί και πέρα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ τους συναδέρφους εδώ και τον κύριο Γούπο και την κυρία Νετσέλεβα για τόσα μας ε, είπαν. Το δίλημα στο οποίο βρίσκεστε αυτό το αντιμετώπισα και εγώ, γιατί ήμουνα και εγώ στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των εκλογών και θυμάμαι πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παρεμφερής με αυτή που περιγράψατε εσείς τώρα. Ε, νομίζω ότι ε, κάπως πρέπει να τα ερμηνεύσουμε και όλα αυτά θετικά. Θυμάμαι ότι όταν μπήκαμε ε, στο εκλογικό τμήμα όπου έπρεπε να μετρηθούν οι ψήφοι, σχεδόν πάθαμε έμφραγμα από βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο μετρούσαν, ε, γινόταν η καταμέτρηση ψήφων. Μιλάμε για το απόλυτο χάος. προσπαθούσαν παραδείγματος χάρη να μετρήσουν ψήφους ε, σε εκλογικά τμήματα που δεν είχαν καν ρεύμα. Μετά το 2006 προσπαθήσαμε να δείξουμε κάποια κατανόηση, ήταν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές, υπήρχαν οι αρχικές ε, δυσκολίες, αλλά ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι μας έμειναν κάποιες αμφιβολίες ε, όσον αφορά στην ε, ικανότητα οργάνωσης σε αυτή τη χώρα. Επίσης ε, διερωτηθήκαμε ε, σε ποιο βαθμό υπάρχουν ε, δόλοι και λατρέοι χειρισμοί. Όλα αυτά δημοσιεύτηκαν, έγιναν γνωστά. Σίγουρα στη χώρα αυτή έχουν γίνει επενδύσεις, αλλά δυστυχώς χωρίς συνέπεια και συνέχεια. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι με βάση τις ε, δικές μας αξίες και αρχές ε, θα παρουσιάσουν την κατάσταση πραγματικά ως έχει. Κυρία Κέλλινης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, αναρωτιέμαι για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ιανουαρίου του 2011, όταν έμαθα ότι τροποποιήθηκε το Σύνταγμα στο Κονγκό. Θέλω να ξέρω δηλαδή, να μάθω, γιατί αποφασίστηκε να επενδύσουμε όλα αυτά τα μέσα και να στείλουμε κόσμο για τις εκλογές στο Κονγκό. Και τι κάναμε σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος. Για άλλε μου ερωτήσει τώρα. Γι' αυτό το σχέδιο νόμου στην Εθνική Συνέλευση, εγώ δεν λέω Δημοκρατία του κογκό, μου έρχεται δύσκολο αυτό το Δημοκρατία στο κογκό. Τέλο πάντων, αυτό το νομοσχέδιο που προέβλεπε ε, να τιμωρείται η ομοφιλοφιλία. Ξέρετε που βρισκόμαστε για αυτό το θέμα, αυτό το νομοσχέδιο διατηρήθηκε ή αποσύρθηκε. Έρχομαι τώρα στη διαμάχη αυτή που πλήττει κυρίως ε, το Ανατολικό Κονγκό. Ξέρουμε ότι τα ορυκτά παράνομα μετακινούνται και βγαίνουν από τη χώρα. Θέλω να ξέρω πώς ε, αντιδρούν οι δυτικές επιχειρήσεις, τι έχουμε κάνει για να τις ευαισθητοποιήσουμε. Υπενθυμίζω ότι ο νόμος του 2010 χαιρετήθηκε από το Κοινοβούλιο αυτό στις 15 ε, Δεκεμβρίου του 2010, όπου συστήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το Αμερικανικό ε, παράδειγμα, πρόκειται για τον Αμερικανικό νόμο, και να υιοθετήσουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο, ώστε να ξέρουμε τα ορυκτά που φτάνουν στην Ευρώπη από πού μας έρχονται ακριβώς. Ελπίζω η Επιτροπή να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο μέτρο το οποίο προτάθηκε για να συνεισφέρουμε στην ε, καταπολέμηση της εισαγωγής ε, τέτοιων ορυκτών από τις περιοχές όπου υπάρχουν οι διαμάχες αυτές. Ξέρουμε ότι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί δραστηριοποιούνται στις χώρες μας. Και ξέρουμε ότι υπάρχει οικονομική στήριξη σε ομάδες όχι και τόσο ειρηνικέ όπως η Φεντέλ και παράδειγμα που δραστηριοποιείται ανατολικά στο Κονγκό. Οι διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δουλεύουν στην περιοχή πολλές φορές έχουν κάνει έκκληση στις δυτικές κυβερνήσεις κυρίως του Βελγίου και της Γαλλίας, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαλύσουν τα δίκτυα αυτά. Θέλω να ξέρω λοιπόν, έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου επί τη ευκαιρία της ε, έκθεσης αυτής που τόσο καλά μας παρουσίασαν οι δύο συνάδελφοι. Ο κύριος Ζέλερ πρώτα να έχει το λόγο και μετά οι συνάδελφοι. Κυρία Νετζέλεβα, παρακαλώ όμως, πρώτα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γίνεται συζήτηση εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την, το σεβασμό μου προς την πρόεδρο της Επιτροπής ε, που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδότησε αυτές τις εκλογές. Το κράτος, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, το προσπάθησε να το κάνει αυτό με τα δικά του κονδύλια. Ε, πάνω από ένα δις λένε ότι κόστησε η όλη ε, προεκλογική εκστρατεία και μάλλον οι εκλογές. Και παρόλα αυτά αποφάσισαν να ψηφίσουν φέτος Ο Νίν, πρόεδρος, πρώην και Νίν, θέλησε να ασκήσει πίεση, το έκανε αυτό σκόπιμα. Εγώ, ε, όσον αφορά τα συναισθήματά μου από αυτή την αποστολή, ε, τα συναισθήματά μου είναι διχασμένα, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα στην Κινσάσα, αλλά πήγα ε, στο, στο στη δυτική επαρχία, μέχρι το Ματάντι, την, ε, το λιμάνι και μου έκανε εντύπωση ότι οι ίδιοι άνθρωποι είχαν πολύ υψηλές φιλοδοξίες σε σχέση με τις εκλογές. Οι άνθρωποι καθόντουσαν σε μεγάλες ουρές με υπομονή μέχρι να μπορέσουν να ψηφίσουν και πολλές φορές αναγκάστηκαν να φύγουν απογοητευμένοι γιατί δεν βρήκαν το όνοματά του στου εκλογικού καταλόγου. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ, η ατμόσφαιρα ήταν ήσυχη. Ε, βέβαια στην ε, επαρχία οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ότι ήταν κατά του Προέδρου Καμπίλα. Ο Ετιέν Τσισεκέντη ήταν ε, ο ευνοούμενός τους. Και στα εκλογικά τμήματα επιτόπου και εκεί διαπιστώσαμε, τουλάχιστον στο Ματάλι, ε, σε μια επαρχία του Κονγκό, εκεί οι τοπικές ε, εφορευτικές επιτροπές προσπάθησαν να ε, οργανώσουν, να διεκπαιρεώσουν σωστά την εκλογική διαδικασία. Και κατά τα άλλα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Σε εμά βλέπω τι στη Γερμανία και πρέπει να σα πω ότι και εγώ μια φορά ήμουνα σε τοπικό επίπεδο υπεύθυνο για την οργάνωση εκλογικής διαδικασίας. Σε εμά λοιπόν πριν από τις εκλογές και την ημέρα των εκλογών υπάρχει κάποια νευρικότητα κατά πόσον θα πάνε τα πράγματα καλά και δύο ημέρες πριν από τις εκλογές είχαμε προσκληθεί στην κεντρική εκλογική επιτροπή, μάλλον τώρα εδώ στο Κονγκό. Είχαμε πάει δύο μέρες πριν, μας ε, κάλεσαν στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και εκεί επικρατούσε άκρα του τάφου σιωπή. Ε, καθόλου ε, αναστάτωση, τα μισά γραφεία ήταν άδεια. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έβλεπε το όλο, την όλη διαδικασία με μεγάλη ψυχραιμία αυτά που ελέγχθησαν περί βίας, ε, πράγματι πιστεύω ότι τελικά η χώρα αυτή δεν θα ερεμίσει και είναι και πολύ μεγάλη σε έκταση για να μπορεί να την κυβερνήσει ένα και μόνο άτομο. Στο Σύνταγμα της Δημοκρατικής, ε, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αναφέρεται ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε ομοσπονδία. Όμως ο πρόεδρος τώρα το διέγραψε, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει, θα προσπαθεί να ε, διοικεί μόνος του τη χώρα, συγκεντρωτικά, κάτι το οποίο Βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν και πολλές φιλετικές συγκρούσεις και πολλές φορές ασκείται βία, εισαγόμενη βία, έρχονται ένοπλες ομάδες, διασκίζουν τα σύνορα, κυρίως βορειοανατολικά και ανατολικά. Εκεί οι πολίτες ε, εκφοβίζονται και τρομοκρατούνται από ε, ένοπλους πολίτες. Αυτό το οποίο απομένει είναι η διπλωματική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών. Αυτοί όμως δεν έχουν και πολλές ελπίδες, δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει γρήγορα η κατάσταση. Κάτι το οποίο βέβαια είναι λυπηρό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι δικό μας καθήκον, καθήκον δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής, είναι δικό μας καθήκον αυτή η χώρα που είναι τόσο μεγάλη όσο μισή Ευρώπη να ε, τραβήξει περισσότερο την προσοχή μας. Παράλληλα, είχαμε εκλογές και στην Αίγυπτο. Αυτές προβλήθηκαν κυρίως ε, στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ε, κανείς σχεδόν δεν ασχολήθηκε με τις εκλογές στο Κονγκό. Νομίζω λοιπόν πολλές από τις καταστάσεις, τις ιδιαίτερα επώδυνες που υπάρχουν στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αυτές ανάγονται το ε, απεικιοκρατικό τους παρελθόν. Άρα δηλαδή φέρουμε και εμείς ευθύνη. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τη χώρα και όπου είναι δυνατό να παρεμβαίνουμε βοηθώντας όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Διότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα ε, παρουσιάστηκαν, αναφέρθηκαν, έχουμε δυσκολίες στην πολιτική δομή, η χώρα είναι διχασμένη, δεν υπάρχει υποδομή. Παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, τουλάχιστον να μην την αφαιρέσουμε από την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Ντελνέτσεβα ε, και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δουλειά που έκαναν. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ντελνέτσεβα ε, αξίζει τις ευχαριστίες μας, κυρίως διότι στις εκθέσεις της και στις γνωμοδοτήσεις της ε, εφαρμόζει δικά μας τα κριτήρια. Δηλαδή δεν πίστηκε ούτε εκφοβίστηκε να μην πει αυτά που είδε ή να τα εξοραίσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι σκάνδαλο και πρέπει να το αναφέρουμε το ότι δηλαδή υπήρξαν τέτοιου είδους προσπάθειες εκφοβισμού. Εγώ πιστεύω ότι το Κονγκό είναι μια χώρα όπου πρέπει κατ' ουσία να πούμε ότι οι εκλογές αυτές ε, με βάση πληροφορίες ε, που είχαμε ε, δεν έπρεπε καν να πάμε να τις παρακολουθήσουμε γιατί ήταν προβλέψιμο ότι δεν επρόκειτο να εφαρμοστούν έστω και οι ελάχιστες προδιαγραφές εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, στις ομάδες εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξαν αρκετοί που είπαν να μην πάμε. Όμως ε, τα κράτη-μέλη άσκησαν πίεση παρόλα αυτά να πάμε. Και είναι πάντα τα ίδια κράτη-μέλη τα οποία αφού εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τώρα θέλουν να τα εξοραίσουν, ε, να τα αθώσουν και να δώσουν μια στρεβλή εικόνα της κατάστασης. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το δεχθούμε στο Κοινοβούλιο. Εγώ στηρίζω 100% τη Μαρία Ντελνέτσεβα όσον αφορά την έκθεσή της και την προσωρινή και το ανακοινωθέν που εξέδωσε μετά την επίσκεψη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε από την Ένωση, από την κάθε Άστον, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Τώρα τουλάχιστον, αφού υποτίθεται ότι το ανώτατο αυτό δικαστήριο ενέκρινε τις εκλογές ε, και τις θεώρησε ανώθευτες, να πούνε τα όργανα της Ένωσης ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ πρόκειται για άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να είναι αποδεκτή, απαράδεκτη πολιτικά. Και εγώ θέλω να γράψω μια επιστολή στην κυρία Άστον και να την καλέσω να ονοματίσει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχω μπροστά μου ένα ε, έγγραφο από την Σένη, από την, ε, που αφορά την Κατάγκα, το εκλογικό τμήμα Μαλαγκουκούλου στις 269.000, από ό,τι φαίνεται, το 99% πήγε, υπήρχε δηλαδή εκλογική συμμετοχή κατά 9% και το 100% ψήφισε για τον Καμπίλα. 100%. Ε, τώρα είναι ντροπή. Ελπίζω αυτό το έγγραφο να μην ευσταθεί, αλλά αυτό που κάνουν που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν, να μας το παρουσιάσει η κυβέρνηση του Κογκό, αυτό είναι παράτολμο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δεχτεί κάτι τέτοιο. Εμείς ε, δεν έχουμε κανένα λόγο να τρέχουμε πίσω από αυτούς τους ανθρώπους με την έννοια να δεχόμαστε τα ψέματά τους που μας αραδιάζουν εδώ. Ακόμα και αν έχουμε οικονομικά συμφέροντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα απαράδεκτα. Εγώ λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι η μέθοδος που θα εφαρμόζεται στην παρακολούθηση εκλογών, αυτή η μέθοδος ε, θα εκφραστεί και στην τελική έκθεση της Μαρία Ντελνέτσεβα. Και ε, θεωρώ επίσης ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφή την πραγματικότητα και περιμένω από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να τα στηρίξουν όλα αυτά, να εξάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα, όχι όπως έγινε ε, το 2006 όπου είπαν η ζωή συνεχίζεται, business as usual. Ευχαριστώ. Μαριά, θέλεις ε, να ξαναπάρεις το λόγο, ναι? Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μας έδωσαν την υποστήριξή τους ε, και την ενθάρρυνσή τους. Είναι αυτός ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Κοινοβούλιο. Βεβαίως δεν έχουμε το ίδιο βάρος στην εξωτερική ε, πολιτική όπως όλη η Ένωση, αλλά είμαστε ένα βήμα που πρέπει να συνεχίσει ε, να λέει δυνατά το τι τα άτομα ε, σκέφτονται στις χώρες αυτές τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Θα ήθελα να επανέλθω σε μερικά σε ερωτήσεις που τέθηκαν για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή της συνταγματική. Να υπενθυμίσω ότι η αλλαγή συνταγματική γίνεται διαμέσου οργάνων που έχουν εκλεγεί και στην περίπτωση της Δημοκρατίας του Κονγκό υπάρχει κοινοβουλευτική συνέλευση. Ποια είναι η νομιμότητά μας αυτού του είδους της αποφάσεις εφόσον λέμε ότι υπάρχουν οργανώσεις που εκλέγονται δημοκρατικά και πρέπει να τηρήσουμε την, την απόφασή τους στην αυθεντικότητα σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό θα επανέρχεται ενώ έχουμε να τηρήσουμε τους διεθνούς κανόνες. Εδώ θα μπορούσα να αντιστρέψω την ερώτηση και να πω πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί αν δεν είχαμε αποστείλει μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως σε σχέση με το 2006 υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή. Η διεθνής κοινότητα έπαιξε εξέχοντα ρόλο. Αυτή τη φορά οι αρχές του Κονγκό ήταν, του Κονγκό ήταν οι κύριοι ε, του παιχνιδιού. Τι ε, μήνυμα θα έστενε το, η Ένωση αν δεν στέλναμε αποστολή. Αντίθετα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι οι αποστολές αυτές υπάρχουν για να γίνεται μια ουδέτερη ανάλυση λεπτομερής της κατάστασης και από εκεί να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή συστάσεις αυτών των αποστολών και ο τρόπο που υλοποιούνται αυτές οι συστάσεις και ποια είναι τα μέσα, οι πιέσεις ακόμα και πολιτικές που μπορούν να ασκηθούν ούτως ώστε οι συστάσεις των αποστολών να μην παραμείνουν νεκρό γράμμα. Υπενθυμίζω ότι οι συστάσεις που έγιναν το 2006, μόνο δύο από αυτές ε, τηρήθηκαν από σημαντικό αριθμό συστάσεων. Από δική μας πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται, να κάνουμε συστάσεις που να είναι ε, ρεαλιστικές, ε, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, να τις διαφοροποιήσουμε, να μην έχουμε τη φιλοδοξία να κάνουμε συστάσεις που ισχύουν για δημοκρατία που έχει μακρά ιστορία, αλλά ε, να έχουμε συστάσεις που να είναι ρεαλιστικές και μετά να έχουμε απέτηση σχετικά με τον νόμο για την ομοφιλοφιλία δεν είναι ρόλος μου, δεν το ξέρω αυτό, αλλά για την κατάσταση ανατολικά του, στα ανατολικά του Κονγκό και εκεί είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγα στον νότιο, νότο και εκεί η εξέλιξη της ασφάλειας της χώρας είναι θετική, εξελίχθηκε θετικά και αυτό χάρη στις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η UPEL, η Αυτές οι αποστολές ε, έχουν τη σημασία διότι μας παραπέμπουν σε δύο θέματα αφενός να εξακολουθήσουμε να αφοπλίζουμε και να καταπολεμούμε τις δυνάμεις, τις στρατιωτικές που παίρνουν τον τρόμο ε, κυρίως ανατολικά και κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει τώρα μια αστυνομία που εκπαιδεύτηκε, καταρτίστηκε, εξοπλίστηκε και που έχει ως εντολή να μην χρησιμοποιεί ποτέ τα όπλα κατά των αμάχων πολιτών και αυτό έχει επιπτώσεις πολύ θετικές και στη συμπεριφορά των αστυνομικών. Το είδαμε την ημέρα των εκλογών ε, μπορέσαν ακόμα και σε μέρες εντάσεως να έχουν μια συμπεριφορά παραδειγματική και βλέπουμε ότι ο πληθυσμός θα πρέπει να θεωρεί τις ε, δυνάμεις ασφαλείας όχι απειλές για την ασφαλειά τους αλλά εγγυητές της τάξης. Ε, σχετικά με το θέμα των ορυκτών. Ε, θα δούμε ε, την μήνα Οκτώβριο. Ξέρουμε ότι η διαδικασία του Κίμπερλε πέτυχε κάποιο συμβιβασμό, ενώ είχε αποτύχει τα πρόσφατα χρόνια θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε ιδέε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγε τι γίνεται με τη διαδικασία του Κίμπερλεϊ, διότι και η Ευρώπη έχει την ευθύνη της σε αυτόν τον τομέα. Άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Περέλο Ροντρίγκε και όλου του συναδέλφου που ήταν παρατηρητέ και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αποφεληθώ της ευκαιρίας αυτής για να συνεχίσω να, υποστηρίζω την καλή συνεργασία ανάμεσα στις αποστολές παρατήρησης εκλογών που βοηθούν την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι η αντιπροσωπεία αυτή είναι αυτή που επιτρέπει την ενίσχυση του πολιτικού βάρους που λείπει πολύ συχνά από διάφορες άλλες αποστολές. Ξέρουμε την κριτική που γίνεται ότι οι αποστολές ασχολούνται πολύ συχνά με τις τεχνικές απόψεις, υπάρχουν εμπειρογνώμενες, αλλά η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντασσόμενο στις αποστολές είναι ένα συμπληρωματικό μέσο για να ενισχύσει το πολιτικό βάρος της Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μαρία. Κύριος Ροντρίγκας. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Η κυρία Νελδετσέβα είπε πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, πτυχές που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ποιος είναι ο ρόλος των παρατηρητών τελικά. Ναι, αλλά όπως είπε και ο κύριος Ζέλερ, υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα αρκετά ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ανακάζεται να μπαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, να τις προλαμβάνει. Και εμείς, αλλά και η διεθνή κοινότητα, γιατί δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί, είναι και οι καναδικές ε, κλπ. Άρα πρέπει να υπάρχει συνοχή και δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή αν ο καθένα κάνει το δικό του. Στι διεθνεί σχέσει. ξέρω ότι μερικέ φορέ η συνοχή είναι δύσκολη, αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να δείξουμε ότι προσπαθούμε να την πετύχουμε αυτή τη συνοχή. Για τη νίκη του Καμπίλα στην Κινσάσα, να σας πω κι εγώ μια ιστορία. Δεν μπορώ να σας πω ποιος κέρδισε, αλλά αν χρησιμεύει σε κάτι, να ξέρετε ότι σε διάφορα εκλογικά κέντρα στην Κινσάσα και σε ένα που είχε 15 εκλογικά κέντρα, σε δύο κέρδισε ο Καβίλα, ενώ στα υπόλοιπα ο Ξεκέλη. Και αυτό συνέβη σε πολλά μέρη, οπότε το 90% μου φαίνεται περίεργο σαν αποτέλεσμα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τόσο μας είπατε που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι, εδώ Ολοκληρώνουμε το σημείο 14. Στα 15 διάφορα δεν έχουμε τίποτα και στο 16 προσεχή συνεδρίαση είναι στις 12 Ιανουαρίου 9 με 12 και 30 εδώ στις Βρυξέλλες. Καλές γιορτές σε όλους σας.